διότι όπως γνωρίζετε αργότερα θα έρθει ανάμεσά μας ο κύριος Γιούνκερ και πρέπει να είμαστε ταυστηρεί με το χρόνο. Για πέντε λεπτά λοιπόν κάθε σκιώδη ηγητής και εν συνεχεία όλοι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Κυρία Μπι Κάνεν, εξ του ΕΛΚ, κυρία Λιν Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αφήστε με να ευχαριστήσω αρχικά την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία της. Δεν πρόκειται να μιλήσω για τα υπέρ και κατά του φόρου, διότι αυτή τη ζήτηση την έχουμε ήδη κάνει. Θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου στην πρόταση και να αναφερθώ σε κάποια σχόλια. Πρώτον, όπως γνωρίζετε, η θέση του ΕΛΚ ήταν υπέρ ενός ε, παρομοιφόρου και εάν ε, αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο. Εμείς είμαστε υπέρ του διεθνούς. Θα πρέπει ως εκ τούτου η Κομισιόν να εργαστεί λίγο πιο ενεργά και αποτελεσματικά στο πλαίσιο του G20 για να έχουμε ένα παγκόσμιο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Γνωρίζω ότι οι συζητήσει που διεξάγονται σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία και άποψή μου είναι ότι ναι μεν ως ομάδα δεν έχουν φασίσει ακόμα, αλλά εάν συμβεί κάτι τέτοιο να υπάρχει ένας ε, φόρος σε θα πρέπει η, Κομισιόν, η Επιτροπή να έχει λόγο και προτείνω ενισχυμένη συνεργασία και το συγκεκριμένο πρότυπο να βασιστεί σε αυτό τον φόρο και όχι επί του τέλους ε, και του χαρτοσύμου. και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις παράπλευρες επιπτώσεις. Κάτι άλλο μας απασχολεί ως ομάδα είναι το ζήτημα των, της έκδοσης ε, Αυτό που μας απασχολεί επίσης είναι και ο ορισμός και τα θέματα αρχής, ε, μιλάω για την αρχή της έκδοσης φυσικά. Επίσης θα θέλαμε να τονιστεί περαιτέρω το θέμα της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. και τις σχέσεις ανάμεσα στις ε, αρχές και τη δυνατότητα κάλυψης τους από ένα ευρύτατο δίκτυο. Αυτά είναι τα κύρια θέματα Επίσης, εάν πρόκειται να εξεταστούν και άλλα εργαλεία, τότε θα πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ κυρία Πιτ Κάνεν. Κυρία Γκουλάρα, εξ τον των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ε, εκ μέρους του Wolf Klins και δι γερμανικά. Ο κύριος Klins καταρχάς ευχαριστεί την κυρία Ποδηματά για την εξαιρετική συνεργασία και θα ήθελα να ρωτήσει τα εξή. Πρώτον, αξίζει να δημιουργηθεί το FTT εάν δεν είναι κανείς στην Ευρωζώνη, εάν δεν εισαχθεί στην Ευρωζώνη ή στην Ευρώ των 27. Δεν θα ήταν καλύτερα μια κοινή λύση. Πόσες χώρες πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα για να αποβεί ωφέλιμο. Δεύτερον, ποιο είδος φορολόγησης είναι δυνατόν μπορούμε ίσως να, να χρησιμοποιήσουμε ως ελάχιστο κατόφλι ε, το stamp duty κατά τα αγγλικά συστήματα. Θα πρέπει, αν επιβληθεί ένας τέτοιος φόρος, να ισχύσει η αρχή της κατοικίας, η αρχή της έδρας ε, και δει σφαιρικά ή πού τέλος πάντων θα επιβληθεί αυτή η φορολογία, αυτό το είδος το stamp duty. Τρίτον, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις ανεπισήμητες ε, επιπτώσεις, παραδείγματος χάρη αυτήν την αλυσίδα επιπτώσεων που θα δημιουργηθεί στο γερμανικό συνταξιδοτικό στο γερμανικό σύστημα Richter ε, το cascading δηλαδή των επιπτώσεων, επιπτώσεις οι οποίες δεν είχαμε προβλέψει. Και όσον αφορά τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, εντάξει, εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε καταρχάς. Και τέλος, τι θα γίνει με τα έσοδα. Ποιος θα, τις, θα συλλέξει τα έσοδα και πού θα, θα διοχετευτούν. Και συνεχίζω στα γαλλικά. Θα ήθελα να πω επίσης ότι το ζήτημα του κριτηρίου της κατοικίας ε, αλλά αυτό ήδη το ανέφερες, ε, πιστεύω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να υπολογίσουμε σωστά και να μην ε, υπάρξει πρόβλημα με την ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω. Ε, ευχαριστώ κυρία Γκουλάρ, εξ των Πρασίνων. Ο Λίγιος Καφέ το Δεδομένου του ότι δεν αντικαθιστώ τον ε, Ανιγκόλ, ε, θα ομιλήσω την γαλλική. Σε ευχαριστώ Άννη για την έκθεση. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία συγκλίνουμε. Να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, ε, σε ό,τι τα δύο τελευταία σημεία συμφωνώ με την Σιλβή. Η χρήση που θα γίνει αυτού του φόρου δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αφορά μόνο τους ίδιους πόρους της Ένωσης. Ε, υπήρξε και μια αρχική βούληση προκειμένου να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος για να χρηματοδοτήσουμε την καταπολέμηση κατά της ένδυας και την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει εν μέρη τουλάχιστον να παραμείνει στον αρχικό στόχο αναφέρεται στην έκθεσή σου και θα καταθέσουμε τροπολογίες και εμείς προς την κατεύθυνση αυτή τώρα το θέμα των συναλλαγών υψηλής συχνότητα. Δεν ε, πιστεύω μάλλον ότι μπορούμε και εδώ να καλθέσουμε τροπολογία, αλλά μπορούμε να προτείνουμε μια διάταξη που θα λέω ότι φορολογούνται ή υποβάλλονται σε φόρο οι συναλλαγές ε, όλων των ε, φορέων που εκδίδουν εντολές και που κατά το μεγαλύτερο μέρος ακυρώνονται διότι το, η ψηλή συχνότητα συναλλαγές έχει ως αποτέλεσμα να περνάνε λίγες εντολές σε σχέση με τον συνολικό αριθμό. Αν καλυφθέσουμε λοιπόν μια τροπολογία για ένα ράσιο, για ένα λόγο, δηλαδή ε, πραγματοποιήσεις ε, συναλλαγές και εναντί ε, των εντολών που εδόθησαν χωρίς να πραγματοποιηθούν θα μπορούσαμε λοιπόν να προβλέψουμε ένα υψηλότερο ποσοστό στο μέτρο που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτή η μορφή της, ε, ε, ε μηχανικής ε, δεν είναι σωστή. Και κάτι ακόμα αναφορικά με το ενδιαφέρον έχουμε τις τρεις αρχές, αρχή της κατοικίας, αρχή της έκδοσης και αρχή της ιδιοκτησίας. Αυτά αναφέρθηκε στην έκθεσή σου, παίρνοντας λοιπόν υπόψη αυτά τα τρία στοιχεία ανάλογα με το προϊόν και την αγορά, θεωρώ ότι μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά το φόρο, τον κίνδυνο φοροδιαφυγής και κάτι άλλο στο οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Συμφωνώ με το όσα είπε παιδικά είναι ότι χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι το ιδανικό είναι να υπάρξει ένας φόρος παγκόσμιος εάν η Ευρώπη θέλει να είναι ηγέτης ε, τότε θα πρέπει να το τονίσουμε. Το, το πλαίσιο όμως της ε, Ευρώπης ε, δεν ξέρω αν θα επιτρέψει σε, να ληφθεί τώρα ένας φόρος σε επίπεδο 27. Αλλά αν δεν ξέρω πότε θα ληφθεί η απόφαση και στην έκθεση της Άνης αναφέρεται ότι κάποια κράτη θα μπορούσαν να πάνε και λίγο παραπέρα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σαφέστεροι και πως ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας στην πολιτική ζήτηση για τον ε, φόρο ήταν ε, να, να σπρώξουμε, να βάλουμε πλάτη για έναν παγκόσμιο φόρο, αλλά αν δεν το κατορθώσουμε τότε πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ξέρουμε ότι το θέμα της ε, νομοθετικής αρμοδιότητας εμπίπτει στα κράτη-μέλη, αλλά χρειάζεται να ζητήσουμε μια καταληκτική ημερομηνία. Εντάξει, η συζήτηση μπορεί να συνεχίσει σε επίπεδο 27 για κάποιε εβδομάδε, μήνε ενδεχόμενα, αλλά μετά θα πρέπει να περάσουμε στην ενισχυμένη συνεργασία. Ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να το μεταθέσουμε για το Σεπτέμβριο, αλλά το Σεπτέμβριο θα είναι καταληκτική ημερομηνία. Από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη θα περάσουν στις ε, ενισχυμένη συνεργασία φυσικά με την τεχνική υποστήριξη της Κομισιόν διότι θα πρέπει να ληφθούν ε, μέτρα τεχνικής φύσης, νομοθετικής φύσης κλπ. για να λάβουμε υπόψη ότι στην ενία αγορά ε, δεν θα παίξουν το παιχνίδι αυτού του φόρου όλα τα κράτη. Εμείς θα κρατήσουμε τροπολογία και να προσπαθήσουμε να πάμε λίγο παραπέρα από ό,τι αναφέρει η έκθεσή σου και να είμαστε πιο σαφείς αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τον χρονισμό της όλης συζήτησης και των αποφάσεων. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω αφορά στην πολιτική επιλογή που έχουμε ενώπιόν μας και πρόκειται για επιλογή ουσίας. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την κυρία Ποδηματά. Θα έλεγα ότι αυτός ο φόρος ε, πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα ως μέσο πίεσης ε, προκειμένου κάποια μέρα να μπορέσει να εφαρμοστεί και σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά Σήμερα ετέθη το ζήτημα αντιστρόφως. Δηλαδή είπαμε ότι θα ίσχυε μόνο εάν εφαρμοστεί παγκοσμίω. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε πρακτικό πνεύμα, από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε χρειάζεται να ξεκινήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτή είναι η προτίμησή μα. Αλλά εάν αυτό πρέπει να το κάνουμε μέσω ενισχυμένη συνεργασία στην ζώνη ευρώ, να το κάνουμε. Αλλά θα ήταν ε, προτιμότερο να εφαρμοστεί σε επίπεδο όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη παρατήρηση. Να πω ότι συμφωνώ με την σχέση ανάμεσα στην αρχή της κατοικίας, αρχή έκδοσης και την αρχή της ιδιοκτησίας στον ΕΛ φόρο αυτόν, την εφαρμογή του φόρου. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους και ήθελα ως εκ τούτου να το αναφέρω και εγώ ρητά. Λοιπόν, ποιες είναι οι αμφιβολίες που έχω. Καταρχήν, ο φόρος αυτός είναι φόρος 0,1% για τις παραδιαστικές συναλλαγές και 0,01% επί των παραγόγων προϊόντων ή τα, πιο, τα πλέον δομημένα παράγωγα υψηλής, για συναλλαγές υψηλής συγνότητας. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σκεπτικό, κάποιος λόγος, κάποιο επιχείρημα πίσω αυτά, διότι αυτό είναι χρήσιμο για τις επενδύσεις που ε, άπτονται στις πραγματικές οικονομίες και προκαλούμε κυρώσεις στις κερδοσκοπικές συναλλαγές. Τώρα, γιατί 0,1 και όχι 0,2 ή 0,3 ε, γιατί το 0,01 και γιατί όχι 0,01 ή 0,03. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάτι τέτοιο. Υπάρχει πολιτικό κριτήριο ενδεχόμενα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε για τον φόρο που επιβάλλει στο νομικό Βασίλειο είναι 0,05 αλλά είχε φτάσει και στο 0,2%. <clears throat> Γιατί λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την Επιτροπή ως αυτού του. Έχω αμφιβολίες επίσης για την αρχή που λέει ότι αυτό θα είναι ένα ελάχιστο και το, τα, κάθε κράτο θα μπορέσει να το εφαρμόσει κάτω δοκούν από εκεί πέρα. Έχω αμφιβολίε, αυτό θα πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό φόρος και όχι ένα διακυβερνητικό. Και εδώ φτάνω στο τρίτο σημείο. Ή αυτός ο φόρος θα είναι ευρωπαϊκός και θα έχει ως αποτέλεσμα ανακατανομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή θα χρησιμεύει αποκλειστικά στις χώρες που έχουν ε, χρηματιστηριακές δραστηριότητες πιο σημαντικές και αυτό δεν ε, είναι απαραίτητο διότι τότε ο, η ανακατανομή θα πλησιάζει το μηδενικό επίπεδο σε επίπεδο χώρας μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα λειτουργεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αναφέρεται τίποτα στην έκθεση. Δεν αναφέρεται τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, σε τι χρησιμεύει αυτό ο φόρο, αν δεν χρησιμεύσει την ανακατανομή, αναδιανομή. Και έχω τελειώσει τον χρόνο που μου δώσατε, κυρία, κύριε Πρόεδρο. Ε, θα πρέπει εδώ να υπάρχει μια άμεση εφαρμογή. Είναι ένας φόρος που εκφύσεις του είναι ένας φόρος αναδυναμητικός. Εάν δεν τον χορηγούμε σε επενδύσεις που αφορούν σε αλλαγές κλίματος, άρα σε μεγάλους στρατηγικούς στόχους της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, τότε θα έχουμε χάσει το τρένο και το ζήτημα αυτό δεν ε, είναι τεχνικό, αλλά είναι καθαρά πολιτικό και που άπτεται της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ κύριε Φούτας. Ε, το γύρο των σκυροδών εισηγητών και περνάμε στους ε, βουλευτές. Σμιτ, Φακούλ, Λούλινγκ και Πιτ Κάνεν. Α, δυσκούλπεν. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ξέχασα τον σκιώδη συγκητή της ε, ε, ομάδας ε, Δημοκρατίας. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την συγκέντρια. Έχω αμφιβολίες όσον αφορά το FTT και για να σας το παρουσιάσω έχω ένα σημείο. Έχουμε έναν τεράστιο κίνδυνο με μικρό απόδοση. Η βασική ιδέα του φόρου δεν ξέρουμε κατά πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό που θέλαμε ήταν να πληρώσουν οι τράπεζες για το κόστος της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δεν νομίζω κατά πόσο αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Ο καταναλωτής δεν είναι εκείνος που θα πληρώσει τελικά, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα ωφέλη από το φόρο αυτό. Παρ' όλα αυτά τα έχουμε τα ωφέλη αυτά ήδη κατά νήμη, ε, Η Κομισιόν υπολογίζει μέχρι και 57 ε, δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι κάπως υπερβολικά αυτά όλα νομίζω. Μια που είναι κάπως απίθανο όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα. Εάν δεν ενταχθούν όλε οι χώρε θα έχουμε στρέβλου συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια αγορά. Λοιπόν, εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιο πολλέ απειλέ παρά ευκαιρίες έχει αυτό ο νέο φόρος. Και αυτή η οδηγία που προσπαθούμε να κάνουμε κατά τι κερδοσκοπίε κατά βάση είναι κερδοσκοπία. Γιατί παίρνουμε υψηλό και, ε, κίνδυνο, αναλαμβάνουμε υψηλό κίνδυνο για μικρό όφελος. Δεν είναι πολύ έξυπνο αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Περκούιτ και με συγχωρείτε που σας, δεν σας είχα δει προηγουμένω. Ο κύριος Ελισσμίθ Σμίθ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Ποδηματά είσαστε μια τολμηρή γυναίκα και ίσως τελικά κερδίζετε, αλλά θα πρέπει να συνεχίσετε να μάχεστε. Δεν είμαι λύση όσον αφορά τους στόχους, τους φόρους, το ξέρετε. Εγώ πληρώνω πολλούς φόρους και μπορώ να το κάνω και ευχαρίστω. Αλλά πρέπει να είναι δίκαιοι οι φόροι αυτοί και θα πρέπει να είναι και ε, καλά δομημένοι και δίκαια δομημένοι. Έχω πολύ έντονες αμφιβολίες ότι αυτός ο φόρος θα το επιτύχει. Θα έλεγα, για να είμαι πιο όμως, ότι είναι κακός αυτός ο φόρος. Άμα θέλουμε να φορολογήσουμε, θα είχαμε νομίζω τη δυνατότητα να ε, πετύχουμε καλύτερη λύση. Παραδείγματο χάρη ένα φόρο FAT ή και VIT, ΦΠΑ. Ε, οι τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και οι διάφορε υπηρεσίε θα πρέπει πραγματικά να συμμετάσχουν περισσότερο. Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και κάπως ρεαλιστές, Πασχάλ. Να μην προσπαθούμε να υπεροβολήσουμε τα πόδια μας, δηλαδή. Έχω δύο ερωτήσεις. Και σχετίστε με αυτό που ε, είπε η Σιλβία ότι είπε ο κύριο Κλίντ πόσες χώρες ή πόσες λίγες χώρες, ποιο είναι το ελάχιστο χωρό δηλαδή που μπορείτε να δεχθείτε. Κάποιος είπε μόνο η Γαλλία και η Γερμανία. Θα ήταν αρκετό αυτό. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Ε, δεν ήξερα αν είσαστε υποψήφια για την προεδρία στη Γαλλία. Δεν πάντων. Είναι σοβαρό το θέμα όμως. Και το άλλο είναι οι ίδιοι πόροι. Η Κομισιόν είπε ότι έτσι μπορούμε να έχουμε κάποιους βιώσιμους ιδίους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είναι όμως μόνο από τους 17 ή και λιγότερους, δεν θα το πετύχουμε αυτό, γιατί κάποιες άλλες χώρες όπως δική μου χώρα, θα πει πρέπει και εμείς κάπου να συμβάλλουμε. Ίσως θα μπορούσατε να μου βρείτε μια απάντηση στις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Σα σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σμιτ. Η κυρία Βόρτμαν Κούλ έχει το λόγο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Άννη για το θαυμάσιο έργο που επιτέλεσε πάνω σε αυτό το γνώμη μου τόσο σημαντικό θέμα. Είναι πολύ αφιλεγόμενο το θέμα, αλλά είναι σωστό ότι το Κοινοβούλιο είναι εκείνο που προωθεί το θέμα και που πρέπει να το προωθήσει. Ακούστηκαν πολλά επιχειρήματα εδώ, με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι με τον φόρο αυτό τον FTT θα μπορούμε να αποφύγουμε μια μελλοντική κρίση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι σαφές ότι και ο χρωματοπιστικός τομέας θα πρέπει να πληρώσει ένα δίκαιο τίμημα όσον αφορά κάποια φορολόγηση. Και μια που προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε ένα πιο βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα, νομίζω ότι εδώ θα είχαμε έναν θετικό ρόλο να δώσουμε σε κάποιες μορφές του FTT. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια πολιτικά, πολιτικές παρατηρήσεις, όχι στο τεχνικό επίπεδο, αλλά στο πολιτικό. Κάποια πράγματα που σκέφτηκα ακούγοντα και διαβάζοντα και τι απαντήσει στην πρόταση τη Κομισιόν, τι γίνεται στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, πώ εκτιμάται η κατάσταση στο Συμβούλιο. Οι προτάσει τη Κομισιόν ε, πολλές φορές οδηγούν σε έντονες αντιδράσεις με καμιά φορά πιστικά επιχειρήματα από την πλευρά των όχι. Κάποια κρατημέλη που δεν είναι, όχι. Υπάρχουν άλλα κρατημέλη που λένε ναι. Εννέα έχουν υπογράψει την επιστολή αυτή. Δεν ξέρω αν τελικά όλοι θα υποστηρίξουν την λόγο πρόταση. Αλλά η πρόθεση είναι ότι ορισμένοι πραγματικά πιστεύουν ότι είναι καλό το FTT, αλλά πολλοί άλλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για τους δικούς τους προϋπολογισμών. Όχι για κλιματολογικές αλληλεγγύες και τέτοια, αλλά πραγματικά για να κλείσουν τα κενά στους δικούς τους προϋπολογισμούς. Για κάποια κρατημέλη και αυτό είναι ένα επιχείρημα, αλλά... Δεν είναι όλοι για αυτή την εναλλακτική που εξετάζει το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να χρησιμοποιηθεί δηλαδή εν μέρη για τον κοινοτικό προπολογισμό. Έτσι δηλαδή να έχουμε επιτέλους ένα τέλος αυτές τις συζητήσει για τους καθαρούς πληρωτές κλπ. κλπ. Αυτά διαβάζω εγώ εν μέρη και στην επιστολή των εννέα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πολιτικά τι θέλουμε. Πολύ φιλόδοξη ε, προσέγγιση όπου 9, 7 ή 6 κρατημένοι εισάγουν ένα FTT ή θέλουμε να προκαλέσουμε και τους 27 με μια πιο βασική αν θέλετε ε, μορφή ε, φορολόγησης με κάποια στοιχεία από το FTT, από το stamp duty της Μεγάλης Δανίας κλπ. Και τι θα έχουμε, θα έχουμε ένα τεράστιο εισόδημα σε λίγα κρατημέλη ή να έχουμε μια πιο ε, απλή προσέγγιση. Εγώ είμαι πάντα υπέρ μιας ε, μέγιστης ε, εναρμόνισης. Εδώ θα είχαμε μια ελάχιστη εναρμόνιση, βέβαια τα κρατημέλη μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα. Αλλά θα ήταν καλό ίσως να προσπαθήσουμε να έχουμε και τους 27 μαζί μας θα άξιζε το κόπο κατά γνώμη μου να εξεταστεί το θέμα στι επόμενε εβδομάδε. σω είναι πολύπλοκο τεχνικά με τι διάφορε τροπολογίε, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια πρόκληση. Εμεί είμαστε πάντα υπέρ τη κοινωτική μεθόδου και η δική μα πρόκληση θα ήταν να προσπαθήσουμε να πείσουμε και 27. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα συνταξιδοτικά ταμεία. Δεν είναι εκείνα αυτά τα οποία πήρανε τους κινδύνους που οδήγησαν στην κρίση και προσπαθούν σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς να κερδίσουν κάποια χρήματα για τις μελλονικές γενιές ε, συναξιούχων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να τους αποκλείσουμε από την οδηγία αυτή νομίζω. Αυτά τα σχόλια και ελπίζω στην Επιτροπή μας ή περαιτέρω να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την απόφαση της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Βάρτμαν Κούλ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να εισαγάγει τον φόρο για τις ε, χρηματοπιστικές συναλλαγές. Αν η Γαλλία θέλει να το κάνει αύριο, αν η Γερμανία ήθελε ήδη να το έχει κάνει από προχθές, θα μπορούσαν να το κάνουνε η συνθήκη το επιτρέπει. Εμείς δεν είμαστε κατά αυτού. Αυτό θα πρέπει να είναι εκ μιας αρχής ξεκάθαρα. Ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να το κάνει αν θέλει. Εγώ θα μπορούσα να έχω μια καλή εικόνα. Είναι ε, ε νομίζω καλό να ε, είναι κανένας ε, φτωχός, ε, οπότε δεν έχω κανένα λόγο να ντρέπομαι. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι παραμένουμε σχολισμένοι στην άποψη του κυρίου Τερεσέ ο οποίος μας προειδοποίησε κατά της εισαγωγής ενός τέτοιου είδους φόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ιδίω βέβαια στην ζώνη ε, ευρώ. Ο κ. Κάκη εξάλλου είχε την ίδια άποψη. Κατά τη γνώμη μου είναι κάπως ε, πολύ νωρίς σήμερα να ε, για το επίπεδο, για το ποσοστό, δηλαδή για την κατανομή των 57 αυτών δισεκατομμυρίων που η συγγήτρια θεωρεί ότι θα είναι το ποσό που θα συλλεχθεί. Όλα αυτά κατά γνώμη μου είναι πολύ πρόωρα. Θα πρέπει πρώτα να ξέρουμε ότι δεν είμαστε ε, κατά του προτύπου, αλλά κατά ε, του ε, παγκοσμίου, ούτε κατά του παγκοσμίου τύπου που θα εισαχθεί στην ομάδα των J20, αλλά όχι εδώ σε μας μονάχα. Καλά τα δώρα, αλλά αυτό πια το ολόκληρο δώρο που πρόκειται να κάνουμε είναι, πώς να σας πω τώρα, ε, παράλογο ας πούμε. Αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για την περίπτωση αυτή, θέλω να πω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ανεπαρκής. Έχει ένα ε, συλλεκτικό διατακτικό Δηλαδή ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται αυξατικά ανάλογα με τον ρυθμό των ε, συναλλαγών στην αγορά. Για ορισμένα χρηματοπιστωτικά ε, προϊόντα, τα, τα μία ας πούμε, τα νιουσίτσφο λέμε που είναι ε, του μεγάλου όγκου στην ευρωπαϊκή αγορά, αυτό θα ήταν ένα θανατηφόρο χτύπημα. Θα πρέπει να πούμε, αν έχουμε να βρούμε ένα διατακτικό, γιατί θα πρέπει να μην ακολουθήσουμε τη γραμμή που υπάρχει εδώ, γιατί θα ήταν απαράδεκτα. Τώρα, εναλλακτική. Δεν θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε μη ένα μόνο φόρο στο χρηματοστήριο. Εάν δηλαδή πράγματι θέλετε μία έκθεση για την πρόταση αυτή της Κομισιόν, στις λεπτομέρειές της, πολλά θα πρέπει να τραποποιήσουμε πάνω στο κείμενο και τις λεπτομέρειες της πρότασης. Καταρχήν όμως είναι σαφής. Σαφές ότι αν δεν εισαχθεί παγκοσμίω θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ επιφυλεκτικοί. Εγώ διασκέδασα λιγάκι με εκείνους που ήδη κατανέμουν τα 57 δισεκατομμύρια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χρηματοδοτικές υπηρεσίες πληρώνουν φόρους 38% του προπολογισμού μας έχουμε από αυτούς. Αλλά εάν τους αφαιρέσουμε κάποια δις ακόμα, θα πρέπει τα εισοδήματά τους να, να φορολογούνται συγγνώμη, λιγότερο. Τι θα γίνει τότε. Και ξέρουμε ότι αυτά τα 57 δισεκατομμύρια, αν μπορούσαν πραγματικά να εισπράξουμε, έχουν δαπανηθεί εδώ τουλάχιστον τέσσερις φορές εδώ στο Κοινοβούλιο και σε κείμενα γραπτά. Πεζολή νομίζω. Θέλει τα χρήματα για την αρτησιακή βοήθεια. Ο κύριος Λάινεν που δεν είναι πια μέλος βέβαια πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος τα ήθελε για το κλίμα. Ο κύριος Λαμασούρ τα θέλει σαν ιδίους πόρους. Ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ τα θέλουν σαν εθνικούς πόρους και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο σφαιρικά και παγκοσμίω, δεν χρειάζεται νομίζω να χρονοτριβούμε με αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούλινγκ για τη τόσο παθιασμένη αυτή η παρέμβασή σας. Η κυρία Μακάρθη έχει το λόγο. Thank you. I mean, I'm probably Ευχαριστώ. Εμείς, εγώ είμαι υπέρ του FTT, εξαρτάται βέβαια τι εννοού, εννοούμε με φόρο στην συναλλαγών. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που αναφέρθηκε σε πολλές πτυχές αυτού του θέματος, ιδίως επί της αρχής του θέματος. Ε, κοιτάξτε, το stamp duty, το χαρτόσημο αυτό που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιτυχημένο. Και είναι επιτυχημένο διότι επιβάλλεται λόγω συγκεκριμένων αρχών. Ένα θεσμικό πλαίσιο ξεκάθαρο. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε αυτό που θέλουμε να επιβάλλουμε έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμο και ξεκάθαρο. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο ε, στη φιλοσοφία αυτής της συζήτησης. Ε, ιδιαίτερα μετά από αυτά που έχουν ελεγχθεί στην ομάδα των συντηρητικών. Εδώ δεν πρόκειται να ξυλοκοπήσουμε τις τράπεζες, να τις δίρουμε. ή θέλουμε να επιβάλλουμε μια πιο θεμητή φορολόγηση και να αποφύγουμε τη φοροδιαφυγή. Εάν κοιτάξετε τι γίνεται φορολογικό καθεστώς μεγάλων εταιριών και πολυεθνικών, δεν πληρώνουν το φόρο που θα έπρεπε ε, χάνονται δισεκατομμύρια από φοροαποφυγή και γι' αυτό αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να εφαρμόσουμε ένα δίκαιο κανόνες του παιχνιδιού και από εδώ και πέρα να πληρώνουν το σωστό φόρο που τους αναλογεί, να συνεισφέρουν δηλαδή δίκαια στο φορολογικό σύστημα. Βεβαίως ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε μια δημοσιονομική κρίση. Ε, αλλά και πιστεύω ότι μπορούμε να ε, δικαιολογήσουμε με θετικά επιχειρήματα την ανάγκη αυτού του φόρου, του FTT. Ε, εν συνεχεία βεβαίως έχουμε άλλες, ε, άλλες ζητήματα να ρυθμίσουμε. Θέλουμε να εφαρμοστεί και στους 27, θέλουμε σε ορισμένους, που και τα λοιπά. Ε, το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε ένα εναρμονισμένο φορολογικό καθεστώς. Αν θέλουμε λοιπόν ομοφωνία ή θα πρέπει να πείσουμε τις χώρες που δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το σύστημα ότι υπάρχουν ωφέλεια θα μπουν και να τους εξηγήσουμε τα πλεονεκτήματα. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι πολλές ε, τράπεζε ε, αισθάνονται μία νευρική ανησυχία. Αλλά Αυτό ε, σημειώστε και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο για την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου. Λένε ότι εμείς μεν θα πληρώσουμε το φόρο, αλλά δεν θα έχουμε δικαίωμα στη μοιρασιά του. Εμείς έχουμε το κοινό σύστημα φορολόγησης μέσω του ΦΠΑ. Ε, εν συνεχεία, ε, το άλλο αντεπιχείρημα ότι είναι μια φορολόγηση υψηλού κινδύνου δεν είναι. Γιατί ήδη το εφαρμόζουν 10 χώρες, αν ήταν επικίνδυνο, γιατί το Χονγκ Κόνγκ το εφαρμόζει ήδη. Το Χονγκ Κόνγκ και άλλες επικράτειες έχουν αυτό το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το ερώτημα είναι όχι τι κάνει άλλη τι κάνουμε εμείς ε, ως ευρωπαϊκή προσέγγιση. Γι' αυτό εγώ συμφωνώ ένθερμα με την πρόταση αυτή και υποστηρίζω τη, τον εισήγητη στη δική μου ομάδα και ε, συμφωνώ με τον κύριο Καλφάν. Αυτό το οποίο δεν θέλω και δεν θα υποστηρίξω, ότι η ομάδα θα το υποστηρίξει, δηλαδή τα μέλη από το Ενωμένο Βασίλειο, και επίσης οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν εκφραστεί πολλές φορές επ' αυτού. Αυτό που δεν θέλουν είναι να χρησιμοποιηθούν ως ε, βούλωμα των ε, ελλείψεων και των κενών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δηλαδή να, τους απο, να απομυζήσουμε ας πούμε αυτούς τους οργανισμούς, τους μη κυβερνητικούς, να τους ε, ρουφήξουμε ας πούμε το φόρο ε, με τη δικαιολογία ότι χρειάζεται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών του κλίματος και των αλλαγών και μετά από 10 χρόνια του πούμε τώρα δεν χρειάζονται η περιβαλλοντική πολιτική αλλά θα συνεχίσουμε να σας ε, αφαιρούμε το φόρο. Δεν πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί ασέμητα και άδικα πρέπει να πείσουμε τον μέγιστο αριθμό κρατών μελών να συνυπογράψουν αυτό το φόρο και να δούμε τι χρήματα θα συλλεχθούν, να δούμε τι ποσά θα συλλεχθούν, εν συνεχεία να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε. Αλλά βασικά ως θεμελιώδης αρχή πιστεύω ότι είναι σωστή επιβολή αυτού του φόρου εν ώψη της οικονομικής κρίσης, της περιβαλλοντικής αλλαγής, ακόμα και της ανεργίας. Η κυρία Τούρνεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Απλώς να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτά που ήδη ελέγχθησαν. Μία ερώτηση προς την Κομισιόν καταρχάς. Είναι εδώ ο εκπρόσωπος, ναι, ωραία. Ένας συνάδελφός σας στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς που είμαι και εγώ μέλος είπε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει πολύ σύντομα μία αναθεωρημένη ή πιο ε, λεπτομερώς μελετημένη άποψη. Μία αξιολόγηση δηλαδή. Πιο λεπτομερή για τις επιπτώσεις αυτού του φόρου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα προσευτεί αυτή η έκθεση που είπατε ότι θα γίνει, διότι πιστεύω ότι οι πληροφορίες από αυτή την έκθεση θα είναι πολύ χρήσιμες, επειδή γίνεται αυτή η έντονη συζήτηση τώρα. Και πολλές χώρες βεβαίως θέλουν να ξέρουν τι επιπτώσεις, τι αποτέλεσμα θα έχει αυτός ο φόρος, διότι οι περισσότερες χώρες είναι σε ύφεση τώρα και σας ρωτώ πότε θα προσευτεί αυτή η έκθεση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη συζήτηση για να ξεκαθαρίσουμε τις απόψεις μας. Δυστυχώς στη Δανία ε, χρησιμοποιήθηκε το χειρότερο σενάριο από την ε, πρώτη έκθεση αξιολόγησης ε, και αυτό είχε μια, έναν αρνητικό αντίκτυπο στη συζήτηση για την όλη οικονομία. Δεύτερον, τα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης. Συμφωνώ με την άλλη Μακάρθη. Κοιτάξτε την, ε, την εμπειρία από την οποία έχουμε ήδη αποκομίσει. 40 χώρες ε, διεθνώς είχαν ή έχουν αυτή τη στιγμή ένα παρόμοιο φόρο. Το μόνο κακό παράδειγμα είναι η Σουηδία. Έχουμε λοιπόν ένα κακό παράδειγμα αλλά και πάρα πολλά καλά παραδείγματα όπου ο, χώρος αυτός, ο φόρος αυτός έχει λειτουργήσει σωστά και έχει βοηθήσει αυτές τις χώρες. Δεύτερον, έγινε μια μεγάλη συζήτηση στην Ολλανδία, η οποία αυτή τη στιγμή ε, γίνεται και στην Δανία, για το συνταξιοδοτικό. Πώς θα επηρεάσει τους συνταξιούχους και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Πιστεύω ότι έγιναν ορισμένες επιθετικές και εχθρικές δηλώσεις στη Δανία ε, από διάφορους που έλεγαν ότι θα πληγούν, θα ζημιωθούν τα συνταξιδετικό ταμεία και συνταξιούχοι. Όμως τα, τα επιχειρήματα αυτά δεν ε, δεν είχαν βάση όπως αντέταξαν άλλοι και δεύτερον, τι άλλα μέτρα μπορούν να εφαρμόσουν οι συνταξιοδοτικά ταμεία, δεδομένου ότι έχουν χάσει τεράστια ποσά κατά την κρίση. Άλλα όμως ταμεία ε, συνταξιοδοτικά έχουν επιβιώσει διότι ήταν πιο σταθερά και πιο μετρημένα στις επενδύσεις τους. Εξαρτάται λοιπόν πώς ε, σχεδιάζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο τα συνταξιοδοτικά ταμεία και εγώ πιστεύω ότι με το φόρο αυτό θα τους ενθαρρύνουμε να επενδύσουν κάπου που είναι ε, οι επενδύσεις πιο σταθερές, πιο σίγουρες. Δεν ε, Νομίζω ε, λοιπόν ότι πρέπει να ακούμε ε, τις, επιθετικές, και εχθρικές απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι γενικά θα είναι ωφέλιμο το αποτέλεσμα. Είπατε και εσείς ότι είσαστε υπέρ του φόρου, δέχεστε να φορολογηθείτε. Εγώ, όπως είπε και η άλλη Μακάρθη, ο φόρος αυτός είναι λογικός, είναι συνετός, θα επιβληθεί σε μια αγορά η οποία παρουσιάζει τεράστια κέρδη και Δεύτερον, όπως λέει και η Κομισιόν, ο τομέας αυτός υποφορολογείται, δεν φορολογείται παρκώς, δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο να αποφύγει την επιβολή αυτού του φόρου που θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη σε αυτή τη φάση που είμαστε. Ευχαριστώ κύριος Μπούλμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε θα δείξω ορισμένα σημεία της συζήτησης. Καταρχάς, η, θέλω να συνεχίσω μετά από αυτά που είπε η κυρία Τουρόνεν και να απευθυνθώ στην Κομισιόν. Πράγματι, από αυτά τα οποία έχει δηλώσει ο αρμόδιος επίτροπος, ξέρω ότι ο ίδιος έχει την εντύπωση ότι οι παλιές μελέτες επιπτώσεων είτε ήταν εσφαλμένες είτε οδήγησαν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Γι' αυτό ακριβώς με ενδιαφέρει ιδιαίτερα πότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια επίκαιρη μελέτη αξιολόγησης, μια καινούρια μελέτη την οποία θα μπορέσουμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε βάσει των τελευταίων συμπερασμάτων. Οι συνάδελφοι οι οποίοι πάντοτε μιλάνε για τη σημασία της εσωτερικής αγοράς, την Ένωση κλπ. κλπ. Αυτούς θέλω να ρωτήσω. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε για φόρους ε, περιορίζεστε στο εθνικό πλαίσιο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη συνάδελφο κυρία Λούλινγκ, η οποία κάθε φορά με κάθε ευκαιρία επενεί την εσωτερική αγορά. Όμως, κάθε φορά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ωφέλη της κοινή αγοράς για την επιβολή μιας κοινή φορολογίας ή φορολογικής προσέγγισης αν θέλετε, τότε αρχίζει και περιορίζεται και αναφέρεται ε, σε εθνικό επίπεδο και όχι ευρωπαϊκό. Ε, ρωτώ λοιπόν όλους, αγαπητοί φίλοι, τι θέλετε να φορολογηθεί εν ώψη της κρίσης που... Θέλετε να φορολογηθεί η εργασία? Θέλετε να φορολογήσουμε ψηλότερο το κόστος εργασίας? Ε, δεν νομίζω. Τι θέλετε. Θέλετε να φορολογήσουμε το, τις, τις επιχειρήσεις, μικρομεσές. Ποιον θέλετε να φορολογήσουμε και πώς. Εάν θέλετε να χειριστούμε αποτελεσματικά την ε, κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αν θέλουμε να παγιωθούν και να συνέλθουν ε, οι προϋπολογισμοί μας, πρέπει να επιβάλλουμε ε, δίκαιη φορολόγηση. Γιατί λοιπόν να μην ωφεληθούν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν θέσεις εργασίας και γιατί να μην φορολογηθούν δίκαια, χωρίς να αποφεύγουν φόρους, αυτοί οι οποίοι ζουν από την κερδοσκοπία και κερδοσκοπικές συναλλαγές. Πολλοί συνάδελφοι λένε, ναι, ναι, εμεί θέλουμε να φορολογηθούν οι χρηματαγορές, αλλά όχι με αυτόν ειδικά το φόρο. Οπότε ρωτώ, στο τέλος της ημέρας, κα, καταλήγουμε, όπως είπε και ο κύριος Σμιτ, καταλήγουμε σε προτάσεις που λένε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τα γκισέ τα, α, τους τελικούς χρήστες, τους τελικούς χρήστες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων χωρίς να τα φορολογούμε τα, τα αφεντικά, χωρίς να φορολογούμε τελικά όλους αυτούς τους έξυπνους οι οποίοι κάνουν τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας ε, χωρίς ε, αυτούς δεν τους φορολογούμε, αυτοί ξεφεύγουν με φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, αλλά φορολογούμε και χτυπάμε κατά κέφαλα όλους τους μικρούς. Με τις μικροσυναλλαγέ, ας πούμε, σε τοπικό επίπεδο, στα γκισέ που γίνονται από ιδιώτες κλπ. Ε, μου θυμίζει αυτό το οποίο λέγεται πολλές φορές το ποδόσφαιρο. Τι ωραίο που είναι το ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο παίζουμε, δεν βάζουμε όμως ποτέ γκολ, άρα να καταργήσουμε το, το δίχτυ του γκολ και να βαράμε όπου θέλουμε. Ε, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη πορεία, συγκεκριμένη δομή. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε αποπροσανατολισμένοι. Ε, πρέπει να ενεργούμε, να δράσουμε ε, και να προλάβουμε τις κρίσεις και το ρίσκο της αγοράς. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ε, υποστηρίζουμε την κυρία Ποδηματά και θέλουμε με μεγάλη πλειοψηφία να περάσει η έκθεση. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούλμαν, ο κύριο Γκαλτιέρη. Ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι η συζήτηση επί του φόρου δημιουργεί ποικίλε αντιδράσεις. Έχουμε και το περίφημο εξώφυλλο του Economist που εμπνέεται από τους βομβαρδισμούς του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου έως ε, τα, την ευχάριστη και την γλαφυρή παρουσία της κυρίας Λούλινγκ. Νομίζω πως ε, και οι δύο αυτές ε, αντιδράσεις είναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι βρίσκονται, μιλάμε για ένα μέσο ε, μπανάλ ε, που δεν θα επιλύσει το πρόβλημα, αλλά αποτελεί έναν φόρο δίκαιο, ισότιμο κλπ. που εξάλλου προϋπήρχε από αρχής χρηματαγορών και χρηματιστηρίων θα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα που έδεσε η συνάδελφος Βόρτμαν Κόλ. Δηλαδή, είπε ο δεδομένου πως ο φόρος θα πρέπει να είναι κοινοτικός, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποκλείσουμε άλλες περιπτώσεις, πιθανότητες και αυτή των ενισχυμένη συνεργασίας, π.χ. διότι έτσι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο το οποίο εμείς θεωρούμε βέλτιστο. Εάν όμως αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα θα μπορούσε να αντιστραφεί ως εξή. Δηλαδή να μην αποκλείσουμε τη δυνατότητα να διανύσουμε άλλες οδούς και μονοπάτια. Θεωρώ ότι από πολιτική σκοπιά είναι ο καλύτερος τρόπος ε, προκειμένου να εφαρμόσουμε ένα φόρο κοινοτικό σε επίπεδο 27. Εάν ε, αποκλειστεί ευθύ εξ αρχή και η δυνατότητα εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό κρατών, τότε το διαπραγματευτικό βάρο σχετικά με την πραγμάτωση αυτού του φόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα είναι εφικτή. Τώρα η πρόταση της Κομισιόν ε, όπως πολύ καλά τροποποιήθηκε από την συνάδελφο Ποδηματά, ειδικά σε ό,τι αφορά την αρχή της έκδοσης, είναι, έχει ως στόχο να τροφοδοτήσει τους ιδίους πόρους της κοινότητας, κάτι το οποίο δεν δικαιολογεί τη συζήτηση που ακούσαμε εδώ από τον συνάδελφο Κάνφιν σχετικά τι θα κάνουμε με, αυτό, με αυτόν τον πόρο. Εάν ε, συμπεριληφθούν στον προπολογισμό της Ένωσης, τότε θα ακολουθηθεί η συνήθις τακτική του προπολογισμού και θα αποφασιστεί η χρήση του. Εμεί σήμερα θα αποφασίσουμε αν πρόκειται να δοθούν στο περιβάλλον, υπέρ τη ειρήνη, τη συνεργασία κλπ. Χρησιμεύουν στο να τροφοδοτήσουν τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει πως... Ε, εάν ε, σε σχέση με ακατανόητα βέτο που ασκηθούν να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος ε, που δεν είναι ο διακυβερνητικός διότι η ενισχυμένη συνεργασία είναι ένα μέσο το οποίο προβλέπεται από τις συνθήκες. Τίποτα δεν ε, εμποδίζει την χρήση αυτών των πόρων τόσο για να αντικαταστήσουμε τις συνεισφορές των κρατών μελών στον προπολογισμό, όσο και μέσω άλλων μορφών που συνδέονται με τις ποικίλε δεσμεύσει που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη της ε, λαμβάνουν στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθεροποίησης ε, και δεν θα ήταν λοιπόν λάθος ε, να νερώσουμε αν θέλετε κάπως την αρχική πρόταση για να γίνει αποδεκτή, αλλά να ενισχύσουμε την πρόταση της Κομισιόν, αλλά ταυτόχρονα να αφήσουμε ανοιχτή και, και το, ανοιχτό και το ενδεχόμενο μιας εφαρμογής του φόρου σε επίπεδο ευρωζώνης. Ευχαριστώ κύριε Καλτιέρη. Η κυρία Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως η συζήτηση αυτή για τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να ειδωθεί σε μια στιγμή όπου το ποσοστό του πλούτου που δημιουργούν οι χρήματα αγορές είναι πιο σημαντικό εδώ και, από ήταν εδώ και 10-15 χρόνια ενώ το ποσοστό του πλούτου που δημιουργείται από την ε, πραγματική αγορά, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά την ε, αμοιβή της εργασίας, έχει μειωθεί και έχει ε, μικρότερα αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πλούτος προέρχεται από τις χρηματαγορές και όχι από την πραγματική οικονομία. Λοιπόν, όταν πρέπει να συνεισφέρουμε, λέει, δεν πρέπει να φορολογήσουμε αυτόν τον πόρο, αυτόν τον πλούτο, συγγνώμη. Αυτό που είναι πιο εύκολο είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο των αμοιβών, το επίπεδο της εργασίας, διότι ε, το κεφάλαιο ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα και συμβάλλει όλο και λιγότερο στην ε, ίσπραξη φόρων και, στα, και στο φορολογικά συστήματα των κρατών μελών. Ενώ λοιπόν διανύουμε μια σοβαρή κρίση και τα κρατη θα πρέπει να χρηματοδοτούν τις ανάγκες ε, των πολιτών, τα κράτη τι κάνουν αντί να επιβάλλουν αυτούς τους, αυτό το είδη των φόρων, επιβάλλουν υψηλότερους ε, φόρους θέμενες αξίες διότι είναι αυτοί οι ε, αυτός ο φόρος ο οποίος ε, μειώνει περαιτέρω το εισόδημα των εργαζομένων δίχως να επηρεάζει την κυκλοφορία των κεφαλαίων. Εάν λοιπόν αυξήσουμε τον ΦΠΑ στο γάλα, στα γαλακτοκομικά, στα τρόφιμα ή την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματο, ε, αυτό τι κάνει, ποιο, ποιος ε, την πληρώνει. Την πληρώνουν οι απλοί πολίτες και όχι όσοι κερδοσκοπούν ε, Λοιπόν, αυτή την, περί... αυτή την περίοδο κρίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε μια επανεξισορρόπηση. Χρειάζεται λοιπόν να επανέλθει η δικαιοσύνη σε ό,τι φορά την ε, συνεισφορά στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών και ζητώντας ε, να επιληθούν πλήρω παραπάνω φόροι σε αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν πρέπει να εξαιρούνται με κανέναν τρόπο, ιδιαίτερα σήμερα. Η επιβολή ενός φόρου σε αυτά τα χρηματιστηριακά προϊόντα είναι κάτι το απαραίτητο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να εξαιρεθούν από την περαιτέρω φορολόγηση στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να καλύψει τις 27 χώρες μέλη. Διότι έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων αλλά και ελεύθερη διακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι στις δυνατότητές μας για να εισπραχθεί αυτός ο φόρος. Ε, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε κατά πόσον, ε, μάλλον πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, αυτοί οι πόροι που θα αποδοθούν Πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα δεδομένου ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει τους ίδιους πόρους της, η σχέση ανάμεσα σε αυτό το νέο εργαλείο χρηματοδότησης και τους ίδιους πόρους της Ένωσης, αυτός ο, αυτός ο σύνδεσμος θα πρέπει να καθοριστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε σε παγκόσμιο επίπεδο να επιβάλλει μια εναρμόνιση, έναν συντονισμό αν θέλετε των πρακτικών που εφαρμόζονται. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε και τον αγώνα μας για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, κάτι το οποίο απασχόλησε και το G20 και σήμερα αυτός ο αγώνας αυτή, κατά των φορολογικών παραδείσων αποκτά ακόμα και μεγαλύτερο νόημα. Θα πρέπει να ξεχαστεί, δεν πρέπει να παραμεληθεί. Η Κομισιόν έχει όλες τις δυνατότητες, έχει όλες τις εξουσίες για να τον επιβάλλει. Εξάλλου ο Σαρκοζή ήταν, ε, έδειξε ιδιαίτερη προνοητικότητα και σήμερα αυτός ο αγώνας, αυτή η μάχη έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από το παρελθόν. Θεωρώ πως η εργασία της κυρίας Ποδηματά αποτελεί μια εξαίρετη συμβολή και ελπίζω πως θα είναι ένας τρόπος για το Ευρωκοινοβούλιο να ανταποκριθεί στα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών και να υποβάλει προτάσεις που είναι πράγματι μοναδικές για την ιστορία μας. Ευχαριστώ. Για μια ακόμη φορά η κυρία Πιτκάνεν έχει το λόγο. Συγγνώμη συνάδελφοι που καταχρώμε το χρόνο σας, αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Πρώτον, νομίζω πως το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι υπέρ αυτής της προτάσεως, διότι τηρεί την κοινοτική μέθοδο, αφορά στα 27 μέλη και συνδέεται με τους ιδίους πόρους σου. Η θέση του ΕΛΚ είναι στεναρός υπέρ των ε, κοινωτικών πόρων και έχουμε αυτή την διπλή θα έλεγα συζήτηση, διότι ξέρουμε ότι συζητήσεις αναφορικά με το χαρτόσημο και τον φόρο επιστηματικών συναλλαγών γίνεται ε, και στο Συμβούλιο και ενδεχόμενα να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία και αυτή η ενισχυμένη συνεργασία σε αυτήν την συνεργασία εμείς δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε ή θα πρέπει να πούμε κάτι τώρα <clears throat> και να υπερασπιστούμε αυτό το σύστημα αλλά εάν προχωρήσει σε επίπεδο μόνο ευρωζώνης ή τουλάχιστον εκτός να μην συμμετάχουν για τα 27 κράτη-μέλη, τι θα γίνει. Το μοντέλο πρέπει να είναι ενιαίο και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να, τον, να εφαρμοστεί το φόρος αυτός είναι ότι αν εφαρμοστούν άλλα μοντέλα όπως το FDT και αυτό ενδεχόμενα να ε, αποτελέσει ένα βάρος, με φορολόγηση μόνο των τραπεζών. Τώρα, εάν πρόκειται για χαρτόσημο, θα πλήξει τις ε, μετοχές ε, και τις άλλες συναλλαγές. Γι' αυτό και απέργευση μας στην Σουηδία. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν η κοινωνική μέθοδος, τότε να εφαρμοστεί μέσω της ενσημείας συνεργασίας. Αλλά αυτό το μοντέλο του φόρου θα πρέπει να αποφασιστεί κάποια στιγμή. Και ε, τι κάνουν, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε γιατί μακρηγορείτε. Έχουμε Ωραία. λιγότερο. Έχουμε λιγότερο από 15 λεπτά. Τέσσερα λεπτά στην Κομισιόν και τα τελευταία 10 λεπτά στην κυρία Ποδήματα. Ας ακούσουμε την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να διαιρέσω την ε, εισήγησή μου σε τέσσερα μέρη. Καταρχάς ε, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την υποστήριξη που έχουμε από αυτή την Επιτροπή γιατί και εμείς προσβλέπουμε στα στοιχεία που θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν την πρόταση της Κομισιόν, τις προτάσεις της Κομισιόν για φόρο φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Ιδίως όσον αφορά τη συμπλήρωση διαφόρων πτυχών της αρχής της έκδοσης και τις ε, προτάσεις για την ε, εφαρμοσιμότητα ε, των άλλων εναλλακτικών ε, λύσεων όπως παραδείγματος χάρη της πρότασης ε, για επιβολή χαρτοσύμου όσον αφορά στις συναλλαγές υψηλής συχνότητας, όσον αφορά το διαχωρισμό επαγγελματιών, χρηματιστών και άλλων χρηματιστών κλπ. κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να απαντήσω καταρχάς την ερώτηση για την έκθεση επιπτώσεων. Εδώ επιβεβαιώνω ότι η Κομισιόν έχει αναθέσει μία έκθεση αξιολόγησης σε εμπειρογνώμονες που θα παρουσιάσει πολλές διευκρινήσεις, πολλές ε, λεπτομέρειες και θα ε, μπορέσει επίσης να διευκρινίσει ερωτήματα τα που έχουν προκύψει επειδή πολλές πτυχές της πρότασης ήταν εκτός πλαισίου, υπήρχαν στεγανά μέσα στην έκθεση και έτσι δεν υπήρχε ένα ενιαίος ε, μια ενιαία συλλογική. Η Κομισιόν πάντοτε θέλει να έχει μια σαφή εικόνα των μακροπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων και για την αγορά εργασίας και για την οικονομική ανάπτυξη. Και ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να ξέρουμε πώς θα γίνει η ανακύκλωση αυτών των εσόδων. Το άλλο θέμα είναι πώς τις επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αυτή τη χυμαρόδη επίπτωση, το cascading impact. Ε, πάντοτε με εκπλήττει το γεγονός ότι ε, δεν ε, μπορεί, μπορεί κάποιος να μεταφέρει την έδρα του ή τις επενδύσεις του εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μεσάζοντες για να ενεργούν εκ μέρους αντισυμβαλόμενων. Ε, υπάρχει μόνο η δυνατότητα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να πληρώσει τους φόρους Εάν ο χρηματιστής και ο μεσάζων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, έχει κάνει άλλες συναλλαγές μεταξύ, μόνο ο τελευταίος αντισυμβαλόμενος θα πληρώσει το φόρο. Αυτή η χυμαρόδη, δηλαδή η αλυσιδωτή αντίδραση η οποία καταλήγει στον τελευταίο φορολογούμενο που θα φορολογηθεί. Ε, όσον αφορά τα συνταξιδετικά ταμεία, έχουμε δει πολλές επικεφαλίδες, πολλούς τίτλους, πολλές κραυγές ε, αρνητικές για τις επιπτώσεις. Όμως πρέπει να διαχωρίσουμε δύο ειδών συνταξιδοτικά ταμεία. Αυτά που ενεργούν συντηρητικά, που δεν θα επηρεαστούν σχεδόν καθόλου μηδαμινά. Και δεύτερον, ε, τα συνταξιδοτικά ταμεία τα οποία ε, θέλουν να αυξήσουν τα, τα έσοδά τους και ε, ε, εφαρμόζουν μια πιο κερδοσκοπική πολιτική. Εκεί ο φόρος που έχει τρία μηδενικά σημεία, τρία κλάσματα μετά το κόμμα, 001 ας πούμε, δεν θα έχει τόσο μεγάλη, δεν θα έχει αυτές τις επιπτώσεις για τις οποίες κραυγάζουν οι αντιτιθέμενοι. Και τέλος, ποιοι θα συμμετάσχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 27 πλην μερικών. Τι εικόνα θα δείξουμε, ότι δεν είμαστε ένα σύνολο, αλλά είμαστε χωρισμένοι σε, σε διάφορες ομαδούλες κρατών. Βεβαίως η Κομισιόν προτιμάει μια σφαιρική λύση, μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία θα είναι καλύτερη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίσης υποβάλει μια πρόταση η οποία στηρίζεται στην προσέγγιση τριπλού α, AAA για όλες τις αγορές που θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη. Όμως, εάν κάποιος ε, θέλει να έχει υπόψη του μια κερδοσκοπική προσέγγιση ή ε, προτείνει κάτι, μια πρωτοβουλία που δεν θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, από τεχνικής άποψης μπορεί να λειτουργήσει βάσει των προτάσεών μας. Απλώς θα μειωθούν θα διαχωριστούν τα κράτη τα οποία εφαρμόζουν το FTT από τα κράτη που δεν τα εφαρμόζουν. Ευχαριστώ πολύ και δίνω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Ποδηματά. Σας είπα 10 λεπτά ή 9 το πολύ, πρέπει να τελειώσουμε. Και ε, θα επικεντρωθώ σε ορισμένα κέρια ερωτήματα. Ε, με δεδομένο ότι ο κ. Μπέρκμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ήδη σε ορισμένα από τα ζητήματα που ετέθησαν. Ξεκινάω από το κυρίαρχο και αιώνιο ερώτημα με το οποίο έκλεισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, εισήγησή της. Ποιο είναι το επιθυμητό ε, επίπεδο για την ε, εισαγωγή αυτού του φόρου, ποιος είναι ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος αντιστοίχως αριθμός κρατών που θα πρέπει να τον υιοθετήσει και να τον εφαρμόσει για να είναι ο φόρος αυτός αποτελεσματικός. θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε κατά νου το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη συζήτηση. Με δεδομένο ότι ε, δεν έχουμε ένα ρόλο συνομοθέτη και άρα με βάση τη δική μας έκθεση μπορούμε να στείλουμε ε, ορισμένα ισχυρά πολιτικά μηνύματα ε, τη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό πολλών κρατών μελών και τη συζήτηση στο εσωτερικό του ε, Συμβουλίου ε, είναι προφανές νομίζω ότι μπορούμε να επαναλάβουμε το αυτονόητο, αυτό που έχει αποτυπωθεί σε ψηφίσματα και σε εκθέσεις που έχουμε υιοθετήσει. Προφανές είναι ότι ε, επαναβεβαιώνουμε τη θέση μας ότι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι επιθυμητό να εισαχθεί σε παγκόσμια κλίμακα στο επίπεδο του G20. Ε, αυτό είναι το ένα δεδομένο, το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε. Το δεύτερο σημείο ε, είναι ότι ε, ως ακριβώς ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση αυτού του φόρου στο επίπεδο των 27 κρατών μελών. Και αυτό είναι επίσης αυτονόητο και δεδομένο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα φτάσουμε στο επίπεδο ενός ευρωπαϊκού φόρου ή ενός παγκόσμιου φόρου και εδώ και αυτή τη λύση αν θέλετε ε, υιοθέτησα και εγώ στο σχέδιο έκθεσης σημειώνοντας ότι αυτές τις προτιμήσεις με τη σειρά που σας τις είπα ε, επαναβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στο global level. Ε, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας για ένα φόρο σε παγκόσμια κλίμακα. Και ταυτοχρόνως, αν θέλετε, αφήνουμε τη δυνατότητα, ενθαρρύνουμε τη δυνατότητα Ενό ορισμένου αριθμού κρατών μελών, με δεδομένο ότι έχουμε ήδη την πρωτοβουλία των εννέα χωρών μελών που έστειλαν τη σχετική επιστολή στη Δανική Προεδρία, ε, να επιταχύνουν ε, την διαδικασία ζητώντας ε, να προχωρήσουν, να προχωρήσει ένας περιορισμένος αριθμός κρατών μελών προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δεδομένο ότι δεν πρόκειται να αποφασίσει, να έχει αποφασιστικό ρόλο ως προς το ποιο είναι ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος αριθμός κρατών μελών ώστε να είναι αποτελεσματικός ο φόρος αυτός, πολιτικά είναι το ορθό να μείνει σε αυτή την προσέγγιση. Το δεύτερο ε, σημείο, σε σχέση με τη διαχείριση των εσόδων, έγινε μια συζήτηση από την οποία προκύπτουν ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο οι διαφορετικές απόψεις, αν θέλετε, και οι διαφορετικές προτεραιότητες. Πάλι όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με δεδομένο ότι η υπόθεση της διαχείρισης των εσόδων δεν θα λυθεί εδώ και δεν θα λυθεί στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, όπως καθίσταται σαφές και από την πρόταση της Επιτροπής, ε, η οποία δεν ακουμπάει στο θέμα της διαχείρισης των εσόδων και ορθώς, για να μην μπει σε ένα ε, ακόμη αμφιλεγόμενο ζήτημα με μεγάλες αντιθέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, αν θέλετε, ε, να επαναβεβαιώσει και ε, γι' αυτό υπέβαλα ορισμένες τροπολογίες ε, κυρίως στα recitals και όχι βεβαίως στα άρθρα τις βασικές του θέσεις όπως έχουν αποτυπωθεί σε προηγούμενα κείμενα και σε προηγούμενα ψηφίσματα και εκθέσεις ότι δηλαδή κάνοντας μία παραπομπή καταρχήν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Medium Term Financial Framework ότι ένα μέρος των εσόδων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Είναι μια συζήτηση όμω που δεν θα γίνει στο πλαίσιο αυτή τη ε, έκθεση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ένα μέρο των εσόδων μπορεί, μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί από του εθνικού προπολογισμού για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλημάτων, για την ανάπτυξη. Δεν θα καθορίσουμε πάλι εμεί με ποιο τρόπο θα γίνει η διαχείριση στο εσωτερικό των κρατών μελών. Και το τρίτο σημείο είναι η επανάληψη πάλι μια βασικών μας θέσεων για την χρήση, ε, για την υποστήριξη ε, πολιτικών κοπών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ναι της κλιματικής ε, αλλαγής ή των στόχων της ανάπτυξης. Τρίτο, το θέμα των συνταξιοδοτικών ταμείων και ολοκληρώνω. Ε, θέλω να υπενθυμίσω τα εξή. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι hedge funds και ότι δεν πρέπει να τα ενθαρρύνουμε να είναι hedge funds. Ε, είναι αλήθεια ε, αυτό που είπαν διάφοροι συνάδελφοι ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία δεν έχουν συμβολή στην κρίση. Είναι όμως εξίσου αλήθεια ότι έχει γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις κακή χρήση των πόρων των συνταξιοδοτικών ταμείων. Για να τα προστατέψουμε πρέπει να τα αποτρέψουμε από επιβλαβείς συναλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο τα αποθέματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Muchísimas Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ποδηματά. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 7η Μαρτίου στι 12 το μεσημέρι. Η εξέραση των τροπολογιών θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί 24 Απριλίου και θα πάμε στη Σύνοδο του Ιουνίου. Παίρνω τώρα στο επόμενο σημείο της μεσαιδιάταξης ε, με την Προεδρία της κυρίας Μπόουλης. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, μερικές ανακοινώσεις πριν συνεχίσουμε. Um, uh, earlier Ησυχία σας παρακαλώ. Νωρίτερα μας ρώτησαν αν μπορούμε να αλλάξουμε την προθεσμία τροπολογιών. Είναι τώρα για το 2 Είναι 12 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Α, ήτανε πέντε και τώρα είναι 12 το μεσημέρι. 12 Μαρτίου το μεσημέρι για το τουπάκ Και θα συζητηθούν οι τροπολογίες μάλλον 26-27 Μαρτίου. Μία εβδομάδα αργότερα. Ε, ενδέχεται να μην υπάρχουν όλες τις μεταφράσεις. Ε, θα προσπαθήσουν θα προσπαθήσει η υπηρεσία, αλλά μία-δύο γλώσσες μπορεί να μην υπάρχουν οι μεταφράσεις. Και εν συνεχεία η ECON ε, θα είναι η συνεδρίαση, δεν θα είναι στις 12 Απριλίου, αλλά θα είναι 24-25 Απριλίου μάλλον. Και έτσι μπορούμε να τηρήσουμε την ίδια προθεσμία για την ECON. και ευχαριστώ ε, τον συμπρόεδρο που με ανακούφισε λίγο στην Προεδρία της Επιτροπής γιατί είχα υπερβολικό φόρτο εργασίας αυτή τη βδομάδα. Προχωρούμε τώρα στο τελευταίο θέμα της υπηρεσίας διάταξης που είναι ο οικονομικός διάλογος. Ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Ευρωομάδας Jean-Claude Juncker. Δεν χρειάζεται ουδεμία παρουσίαση του κυρίου Γιούγκερ, ε, τον ξέρετε, σίγουρα είσαστε ενήμεροι για τα υψίστη σημασία, ε, τις της σημασίας εξελίξεις που έχουν σημειωθεί πρόσφατα και θα του δώσω το λόγο τα πρώτα δέκα λεπτά ε, για να μας ενημερώσει και εν συνεχεία θα έχουμε ερωταπαντήσεις βεβαίω. Θα ήθελα επίσης να πω στα μέλη ότι υπάρχει μια συνέντευξη μετά δεν μπορείτε λοιπόν να τρέξετε όλοι να τον περιτριγυρίσετε και να τον απομονώσετε έξω από την αίθουσα διότι υπάρχει συνέντευξη τύπου αμέσως μετά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ε, πως δεν έχουμε το απαραίτητο χρόνο για να επεκταθούμε στο ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα, διότι μετά αυτή τη συνεδρία και μετά από το Press Point θα συναντήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και επιθυμώ να μπορέσω να τους αφιερώσω τον ε, απαραίτητο χρόνο διότι η εκπρόσωποι των μισθετών είναι πρόσωπα τα οποία εκτιμώ ιδιαίτερα και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θέσεις τους. Θα ήθελα εντάχει να διαπτέξω τα διάφορα σημεία που απασχολούν τόσο τις εργασίες όσο και αυτές της ευρωομάδας χωρίς όμως ε, να ε, δείξω αναλυτικά την μία ή την άλλη πτυχή εκφραζόμενος ε, με τρόπο, θα έλεγα, περίπου τηλεγραφικό. Θα ήθελα πρωτίστως να αναφερθώ στο ελληνικό ζήτημα, το ελληνικό πρόβλημα. Γνωρίζετε πως στις 20 Φεβρουαρίου και ε, στις 21 ε, θυμάμαι πότε ήταν καθ' τη διάρκεια του πρωινού ε, το Eurogroup μπόρεσε να λάβει μια απόφαση που αφορά ζητήματα αρχής επί του δεύτερου προγράμματος βοήθειας της Ελλάδας που αφορά τα 130 δις ευρώ, τον οποίο ο διτός στόχος είναι να διασφαλίσει την ε, στήριξη του ελληνικού χρέους και να προωθήσει την αραγωνιστικότητα της χώρας η οποία υποφέρει από απώλεια της αραγωνιστικότητας μετά από την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Συμφωνήσαμε σχετικά με μια συνεισφορά του ιδιωτικού κλάδου, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν, άγνωστο μέχρι τώρα στην Ευρώπη ο ιδιωτικός τομέας ε, θα αφορά τον ε, κούρεμα 53,5% του χρέους. Θα, θα γνωρίζετε ότι η απόφαση της 26 Οκτωβρίου του Συμβουλίου συμφώνησε για την εθελοντική ε, συμμετοχή του ιδρύου κλάδου κατά 50% στο, στο πλαίσιο των νυχτερινών συζητήσεων προσπαθήσαμε να αυξήσουμε περαιτέρω την το ποσοστό αυτό στο 53,5% κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα αποβεί εις βάρος του ιδιωτικού κλάδου. Το, το συνολική συμμετοχή του ενδέχεται να φτάσει και το 70% στόχος της όλης προσπάθειας, όλου εγχειρήματος ήταν ε, να συνδυάσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού κλάδου αλλά και μια περαιτέρω συμμετοχή του δημόσιου κλάδου για να οδηγηθεί το ελληνικό χρέος μέχρι το 2020 σε 120,5% του Ε, μια μείωση κατά τη ε, μεγαλύτερη αυτή που είχε αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Οκτώβριο. Ε, ξεκινούμε λοιπόν ε, τι διορθωτικές δράσεις με με μία μείωση 129% όπως είχε προβληθεί αρκετά και σιγά σιγά προοδευτικά μπορούσαμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό από 129% σε 120,5% του ΑΕΠ ως το 12 το PSI ξεκίνησε στις 24 ε, Φεβρουαρίου και θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα κατά γύρω στις 9 Μαρτίου ενεστώντος έτους το ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να είναι υψηλό, θα πρέπει να φτάσει στο 66% έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε περαιτέρω και θέλω να καλέσω τον ιδιωτικό τομέα να αντιδράσει με θετικό τρόπο στην πρόταση που τους έχει γίνει. Αυτό θα διευκολύνει σημαντικά την πρόοδο των διαφόρων φάσεων για το συνολικό διάβημα που αφορά το ζήτημα της Ελλάδας. Όταν τα αποτελέσματα του PSI γνωστοποιηθούν, θα προχωρήσουμε σε μια απόφαση αναφορικά με το private sector involvement, τη συμμετοχή του ειδικού κλάδου και θα επισημοποιήσουμε τη συμφωνία μετατρέποντα σε απόφαση που θα αφορά το δεύτερο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα. Το Eurogroup θα το πράξει αυτό γύρω στις 12, 13 με 14 Μαρτίου. Έχουμε συγκαλέσει για αύριο στις 2 ε, το μεσημέρι μια άλλη συνεδρίαση του Eurogroup, κατά τη διάρκεια της οποίας ε, οι Έλληνες συνάδελφοι θα μας ενημερώσουν ε, επί της διεξαγωγής της όλης επιχείρησης, τη συμμετοχή του ιδιωτικού κλάδου. Θα ελέγξουμε κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο έλαβαν Αποφάσει ε, νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με τις προτεραιότητε ε, τι οποίε καθορίσαμε κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεω ε, τη 20 Φεβρουαρίου. Η Ελληνική Βουλή και η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει εισαγάγει ή και εγκρίνει τις κατά προτεραιότητα δράσεις προτού να λάβουμε απόφαση επί του δευτέρου προγράμματος που υποβάλλεται σε κάποιες προϋποθέσεις και την πλήρωση ορισμένων συνθήκων και όλα αυτά αποτελούν ε, μέρος ε, των όρων ε, που εμπίπτουν στο δεύτερο πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν στο σύνολό τους τις αποφάσεις επί των οποίων συμφωνήσαμε γνωρίζετε πως ε, στο παρελθόν οι ελληνικές αρχές δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε όλες τις ανησυχίες μας, αλλά είμαι πεπισμένος ότι μετά από τόσο καιρό και από τόσες ε, ε, παιδαγωγική ε, φύσης σχέσης με την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να ικανοποιήσει ε, τα αιτήματά μας, ε, κάτι το οποίο δέχθηκαν διότι ήμασταν σε θέση να συλλέξουμε, να πάρουμε μάλλον τις υπογραφές των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων, δύο μεγάλων πολιτικών οικογενειών που αποτελούν και τον κυβερνητικό συνασπισμό. Αλλά όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ε, εντάχει μέχρι τα μέσα Μαΐ, Μαρτίου, διότι η πρώτη δόση θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο στις 20 Μαρτίου προς την Ελλάδα. Δεν θέλησαμε λοιπόν να... Ε, αυτό που θέλαμε ήταν ε, να βοηθήσουμε την Ελλάδα και όχι να την ταπεινώσουμε, να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς και να θέσουμε στην διάθεση της Task Force επιπλέον ε, πόρους και να συμπεριλάβουμε στου εμπειρογνώμονες τη Τρόικα και εθνικού εμπειρογνώμονες που προέρχονται από διάφορα κράτη-μέλη τη Ένωση, να ενισχύσουμε τι διοικητικέ αρμοδιότητε και ικανότητε τη Ελλάδα, διότι δεν είναι πάντα οι κατάλληλε. αυτό ότι μια διοικητική αρρωγή, μια διοικητική συνδρομή ουσιαστική φύση είναι απαραίτητη για να εξοπλίσουμε τι ελληνικέ αρχέ, την ελληνική διοίκηση να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις ε, που έχει. Θα... Δεν έχουμε καθορίσει ακόμα όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον ειδικό λογαριασμό, ο οποίος θα επιτρέπει στην Ελλάδα να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους κάτι το οποίο θα συμπεριληφθεί και στην Εθνική Νομοθεσία της Ελλάδας, αλλά και θα εγγραφεί στο Ελληνικό Σύνταγμα. Αυτά σε ό,τι φορά την Ελλάδα. Αλλά δεν είναι, το, δεν τα πάντα αυτά, διότι για μια ακόμη φορά θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι πρέπει να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε το δημοσιονομικά της Ελλάδας, δίχως ε, κατάλληλα ε, κατά τη δημοσιονομική πολιτική, δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το έλλειμμα, δεν μπορούμε να αθρίζουμε και ε, χρέος επί χρέους, σε, ειδικά σε ένα έλλειμμα όταν αυτό είναι υψηλό. Η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στον ελληνικό λαό και στην Ελλάδα, όταν ο, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας υποφέρει πολύ, δεν είναι να επαναλαμβάνουμε από το πρωί στο βράδυ μέρα με τη μέρα να κάνουν οικονομίες και να περικοπές στον προπολογισμό. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τον πιο λογικό τρόπο, αλλά είναι προφανές πως μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα θα πρέπει να υλοποιηθεί. Και αυτές τις μέρες θα το συζητήσουμε το θέμα, στα, σε επόμενες συναντήσεις μας ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κινητοποιήσουμε ε, οικονομικά και χρηματοδοτικά αλλά και τεχνικά μέσα προκειμένου να ε, την ε, ελληνική ανάπτυξη και η πολιτική δεν ε, συνοψίζεται μόνο με την επιβολή κάποιων κυρώσεων και μέτρων τα οποία είναι ιδιαίτερα ε, επώδυνα για τον ελληνικό λαό, αλλά για την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα στοχεύουν στην ε, ανάπτυξη, στη μεγένθηση και να πω επίσης, κυρία Πρόεδρε, μερικά πράγματα επί του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ε, εφαρμογή του οποίου κατέστη δυνατόν από την υπογραφή της συνθήκης στις 2 Φεβρουαρίου 2012 θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2012, διότι αποφασίσαμε να προτάξουμε την θέση ισχύ του μηχανισμού, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, το FSF, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα προγράμματα, τα εφιστάμενα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης, δηλαδή ο μηχανισμός ο οποίος ε, ε, εφαρμόζεται τώρα θα μπορεί να λειτουργήσει πλέον μετά από τον Ευρωπαϊκό, με τη θέση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Το Ευρωκοινοβούλιο φυσικά θα ενημερωθεί για τον τρόπο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, εφαρμογή και λεπτομέρειες επί των οποίων εργάζεται ο κύριος Κλάουδ Ρέγκλινγκ, ο οποίος ε, ε, των οποίων συνδράμουν ε, σημαντικοί εμπειρογνώμονες, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό. Ε, οι εργασίες όμως προχωρούν με γοργό βήμα και θα σας ενημερώσουμε για την εφαρμογή του μηχανισμού και τις δραστηριότητες αυτού. Η συνθήκη γνωρίζω ότι δεν το προβλέπει για λόγους διακυβερνητικούς που γνωρίζετε, διότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεν έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη, αλλά ε, ο πρόεδρος του Eurogroup είναι προφανές ε, πως θα σας ε, ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα αυτό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και την υλοποίησή του τώρα σε ό,τι αφορά την ικανότητα του FSF και του μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας θα πρέπει να διακρίσουμε τις φάσεις ε, και τα διακυβεύματα από τον 1η Ιουλίου 2012, δηλαδή μεταξύ Ιουλίου 2012 και ε, Ιουλίου 2013 η συνολική δυνατότητα του ε, μηχανισμού σταθερότητας θα ανέρθει σε 500 δις και έχουμε αποφασίσει τον Οκτώβριο αν δεν κάνω λάθος τον Ιανουάριο που επαναλαμβάνονται τα συμβούλια το ένα μετά το άλλο θα διάρκεια αυτών των ενός των δύο συμβουλίων θα κυρωθούν αυτές οι αποφάσεις. Δεν ξέρω πότε λάβαμε την απόφαση, αλλά τόσο αποφασίσαμε να επανεξετάσουμε τον Μάρτιο το συνολικό ποσό του μηχανισμού σταθερότητας ε, Είχα σκεφτεί πως αυτή η αναθεώρηση θα μπορούσε να γίνει κατά από κατάλληλες συνθήκες ε, στο αυριανή ή μεθαυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν διότι ε, όλος ο προβληματισμός στις κυβερνήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και εκτιμώ πως πρώτον θα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα της ε, επιχείρησης PSI, να παρθέψουμε αν μέχρι τότε η Ελλάδα θα πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε, που της έχουν ζητηθεί ή μάλλον που έχει η ίδια θέση τον εαυτό της προκειμένου να περάσουμε στην αξιολόγηση του ε, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας να πω ότι η πραγματική ικανότητα θα εξαρτηθεί από την ε, ρυθμό πληρωμής του κεφαλαίου που θα έχει απελευθερωθεί, αποδεσμευθεί. Ε, στο Eurogroup είχαμε αποφασίσει πριν από μερικούς μήνες πως ε, το κεφάλαιο που θα αποδεσμευόταν θα καταβαλόταν σε μία δόση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως μερικές μέρες αργότερα αποφάσισε να καταβληθεί σε πέντε δόσεις ε, αυτό το κεφάλαιο που θα έχει αποδεσμευτεί. Είναι προφανές ότι η κλιμάκωση σε πέντε δόσεις θα σήμαινε μια προσέγγιση πολύ επιφυλακτική, πολύ μετριοβαθή. Γι' αυτό ετοιμαζόμαστε να λάβουμε μία απόφαση προκειμένου να επιταχύνουμε την αριθμό της πληρωμής, της καταβολής και έχω βάσιμους λόγους να πιστεύω ότι το αποδεσμευθέν κεφάλαιο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις και αυτό έχει τη σημασία του στο μέτρο που κάθε δόση αυξάνει την ικανότητα του μηχανισμού σταθερότητας κατά 100 δις. Λοιπόν, εάν θέλουμε να δώσουμε όθηση μεγαλύτερη στον μηχανισμό σταθερότητας θα πρέπει να φροντίσουμε το αποδεσμευτικό κεφάλαιο να καταβληθεί σύντομα και θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στην επιτάχυση αυτής της καταβολής του αποδεσμευμένου κεφαλαίου. Μέχρι τώρα όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμφωνήσει για τη συμμετοχή αυτή στην ε, επιταχυνημένη καταβολή, αλλά Πιστεύω πως ε, εντός ολίγου θα λαβηθεί η απόφαση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε. Προσωπικά κρίνω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε το EFSF και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να αυξήσουμε την ε, ικανότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, και η υπέρ μεταφοράς των 40 δις που θα χρησιμοποιηθεί προς τον, από το EFSF στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας έχοντας κατά νου πως οι διεθνείς μας ε, εταίροι μας ζητούν έντονα και με τρόπο ελάχιστα διπλωματικό να αναλάβουμε κάθε πρωτοβουλία που ενδέχεται να ενισχύσει το τείχος προστασίας ε, που θα αποτελέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Ε, και τώρα τάχει Σάρων ε, να αναφερθώ στην πρόληψη και τη διόρθωση των ανισορροπιών λόγω υπερβολικού ελλείμματος Υπάρχουν κάποιες ε, καινοτομίες ε, στο μηχανισμό οικονομικής διακυβέρνησης. Θα είδατε, όπως και εγώ, ότι στην, ε, η Κομισιόν στην εκθεσή της αποχώρησε στην Eurogroup κάποιες χώρες που χρειάζονται πιο έντονη έργο. Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Βε... ε... Φιλανδία και κάποιες άλλες χώρες θα εξετάσουμε τις σχετικές εκθέσεις στην Ευρωγκρουπ στις συνεδρίασεις 12 και 13 Μαρτίου όσον αφορά την δεύτερη δεσμή της διακυβέρνησης, του διοκονισμού, δηλαδή που είχε υποβάλει στο φθινόπωρο στο Κοινοβούλιο Κομισιόν. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις να κάνω. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η Δανική Προεδρία θέλει οριστικά με το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει την υιοθέτηση των δύο αυτοκανονισμών το καλοκαίρι του 2012. Ξέρω εδώ ότι η συγκεκριτή σας εργάζεται σκληρά πάνω σε αυτούς τους δύο κανονισμούς και από ό,τι ξέρω η Επιτροπή σας έχει προβλέψει να το εξετάσει σχεδόν ολιστικά μέσα Απριλίου αυτό είναι ένα θέμα που εξαρτάται από το Συμβούλιο Εκοφθήνα. Δεν προχωρά λοιπόν ιδιαίτερα γρήγορα, αλλά ε, μια που αφορούνται κυρίως οι χώρες ε, της ζώνης ευρώ, θα είμαι έτοιμος να ακούσω τα πρώτα σας συμπεράσματα πάνω σε ένα κείμενο που είναι αρκετά προβληματικό όπως ξέρω. Δύο λόγια την Ιρλανδία, κυρία Πρόεδρε. Μόλι ενημερωθήκαμε χθε το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό Υπουργό Οικονομικών τη Ιρλανδία για το ότι κατόπιν της σύσταση γνωμοδότησης θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Η Ιρλανδία δηλαδή θα χρειαστεί να περάσει σε δημοψήφισμα για τα αποτελέσματα της ε, οικονομικής ε, σύμβασης. Θα πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή των Ιρλανδών. Οι δημοκρατικές διαδικασίες της Ιρλανδίας είναι αυτές που ξέρουμε. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε αγενείς παρατηρήσεις ε, εν της Ιρλανδίας. Υπάρχουν ορισμένε βουλές στην Ευρώπη και μέσα στην Ευρωζώνη ομάδα στο Eurogroup ε, όπου οι διαδικασίε τους είναι πολύ πιο πολύπλοκες από ότι άλλων. Δεν θα πρέπει να επικρίνουμε την Ιρλανδία για την επιλογή αυτή, κάνοντας τους έξυπνους. Ε, δεν θα γίνει γλίγορα φαντάζομαι αυτή η... αυτό το δημοψήφισμα γιατί χρειάζεται καλή προετοιμασία ο Υπουργός Οικονομικών θα μας ενημερώσει φαντάζομαι ε, γέρα στην Ευρωγκρούπ, αλλιώς θα το κάνει ο Πρωθυπουργό την Πέμπτη το βράδυ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα πρέπει βέβαια να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια γέφυρα μεταξύ της ηθίκης αυτής και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, και η ε, συνθήκη αυτή η οικονομική θα τεθεί σε ισχύ μετά που θα επικαιρωθεί από 12 κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν ερωτηματικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον η Ιρλανδία μπορεί να στραφεί προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για συμπληρωματική ευρωπαϊκή βοήθεια εφόσον δεν έχει ε, εγκριθεί η σύμβαση μέσω του δημοψηφίσματος. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επιμένουμε ιδιαίτερα στη δυσκολία αυτή. Αυτά. Κοιτάξτε τι λέει το κατηχητικό της ε, Καθολικής Εκκλησίας. Λέει στο πιο πικρό το τμήμα. στο πώς ε, μπορείτε να αποδείξετε ε, την ύπαρξη του Θεού δίνει μια πολύ απλή ερώτηση. Αυτό το θέμα δεν τίθεται. Ε, το ίδιο ισχύει και για το θέμα που έθιξα μόλις τώρα. Σήμερα συζητείτε το θέμα αυτό χωρίς ε, και αναρωτιόμαστε περισσότερο για το τρίτο πρόγραμμα της Ελλάδα, από ότι για το δεύτερο πρόγραμμα της, για την Ελλάδα. Ας εφαρμόσουμε το δεύτερο πρόγραμμα για την Ελλάδα, φαντάζομαι με καλούς όρους, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό και να μην κατηγορούμε τον ελληνικό λαό για κάποιες κακές προθέσεις. Ας φροντίσουμε να βοηθήσουμε τους φίλους Έλληνες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και α συγκεντρώσουμε την προσοχή μας από εδώ και μπρό στη πολιτική ανάπτυξη που πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να, να συμπληρώσει τις ε, ε, οικονομικές προσπάθειες της Ελλάδας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε κάθε φορά που σας είσαστε εδώ μαζί μας και βλέπω ότι μιλάτε ελεύθερα, δεδομένου ότι έχετε μόνο μερικές σημειώσεις σε ένα ε, χαρτί από το ξενοδοχείο Σοφιτέλ. Ε, δεν έχετε δηλαδή ένα προετοιμασμένο λόγο, τον οποίο ετοίμασαν οι βοηθοί σα ε, και έτσι μας εκφράζετε τη σκέψη σας με έναν πάρα πολύ ρεαλιστικό και ανθρώπινο τρόπο και ε, έχουμε πολλά ε, θέματα να σας ρωτήσουμε. Σήξατε κι εσείς ε, πολλά σημεία. Uh, so... Και 15 λεπτό είναι ο χρόνος ομιλίας σας. Κα, καταρχάς θέλω να δώσω το λόγο στις ομάδες. Ponimata, Roberto Galtieri, Philippe Lamberts and Nicholas Shuntis. If there's anybody else... Uh... Τελευταία ήταν ο κύριος Χουντής. Okay, I'm, I'm going to close the list at that. Και ε, ολοκληρώνω τον κατάλογο των ομιλητών. Καταρχάς, ο, ο κύριος Τζον Φόρ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είσαστε ένας από τους σπάνιους πολιτικούς ε, της Ευρώπης που έχουν το μειονέκτημα να μιλάνε και ειλικρινά και με σαφήνεια μειονέκτημα λέω γιατί άλλοι θα το αισθανόντουσαν ίσως ε, για κάτι αρνητικό. Καμιά φορά εδώ μαθαίνουμε αυτά που την προηγούμενη είχαμε διαβάσει στην εφημερίδα. Με εσά σώμα σήμερα έμαθα ότι δεν είχα διαβάσει σωστά την εφημερίδα. Είχα την εντύπωση ότι το θένομα της Ελλάδας είχε διακανονιστεί. Αυτή ήταν η τίτλη τυχαίοι που έδωσαν οι εφημερίδες ε, στους ε, πολίτες σώθηκε ο ελληνικό λαό, θα είναι ήσυχοι για δύο χρόνια, είπαν οι πιο αισιόδοξοι. Τώρα όμω ακούω ότι όλα ακόμα βρίσκονται εν ροή. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν που δεν έχουν γίνει ακόμα και βέβαια συμμερίζω με την άποψή σα ότι δεν πρέπει να ταπεινώσουμε τον ελληνικό λαό και θα πρέπει και κάποια στιγμή να ανοιχτούν οι υποχρεώσεις και να έχουμε εμπιστοσύνη η Ευρώπη πρέπει να είναι μια κοινωνία εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις προφορές που μας δώσατε. Ελπίζω οι Εφημερίδε να προέτρεξαν ε, για άλλη μια φορά τον ε, τίτλο που θα πρέπει να έχουν σε μερικές ημέρες όταν θα έχουν ε, επιληθεί όλα τα προβλήματα. Αναφερθήκατε στου δύο κανονισμού που υπάρχουν επιτάπητος κύριε Πρόεδρο. Η κυρία Φεραίρα είναι η συγκίτρια τη μία, εγώ για την άλλη έκθεση. Έχουμε μία πρόταση να κάνουμε που λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των χωρών εν κινδύνο. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε αυτήν την απλοϊκή άποψη ότι αυτό που έγινε στην Ελλάδα θα ήταν απολύτως αδύνατο ποτέ τον ποτό να συμβεί κάπου αλλού. Και γι' αυτό είναι καλό να υπάρχει ένα νομικό καθεστώς για την προστασία των χωρών που βρίσκονται σε δυσκολίες που να βασίζεται στην κατάσταση και τα καθεστώτα που υπάρχουν για τις ε, ε επιχειρήσεις και δυσκολίες ε, όπως παραδείγματο χάνει στη ΣΥΠΑ με το Chapter 11, το κεφάλαιο 11. Γιατί αναφέρεται μια κάποια κατάσταση συγκεκριμένη, είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει ένα ξεκάθαρο καθεστώς να ξέρει ποια είναι η θέση του συμπληρωμένων και των πιστωτών του μια χώρα, παρά να παραμένουν όλα έτσι σε ασάφια και λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σωτηρία τη τελευταία στιγμή, σε μια διάσκεψη κορυφή τη τελευταία στιγμή, κλπ. Και την επόμενη φορά πάλι ξαναρχίζουμε. σα εύχομαι λοιπόν πολύ κουράγιο κύριε Πρόεδρε και οπωσδήποτε έχετε την υποστήριξή μα. If you want to reply, he's left you a minute. Θέλετε να απαντήσετε. Ένα ένα λεπτό σας άφησα. Περίσευμα. ναι. Δεν θέλω να πω στον Ζωπόλ ότι επί του ουσίας, ε, οι ε, ανακοινώσει του τύπου ήταν σωστές. Δηλαδή το δεύτερο πρόγραμμα για την Ελλάδα υιοθετήθηκε. Καταρχήν. Και είμαι αναγκασμένος να σας πω νομίζω εδώ ποια είναι τα άλλα στάδια τα άλλα στοιχεία της που θα πρέπει να τύχουν βασμό. Γιατί αποφασίσαμε να υπάρχει ένα σύστημα πιο αυστηρής και στενής εποπτείας και θα πρέπει να ελέγχουμε κατά πόσον οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία ή όχι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χρηματοπιστός τομέας θα δώσει 170 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και επίσης ζητήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση που συμφώνησε με αυτό ότι θα υπάρχουν ορισμένε δράσει προτεραιότητα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Και προτού ληφθεί μια νομική, αν θέλετε, απόφαση για το δεύτερο πρόγραμμα, χρειάστηκε να ελέγξουμε κατά πόσον αυτέ οι ε, πράξεις προτεραιότητας, ε, τις οποίες έχουμε δώσει με κατάλογο στην ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε δημιουργήσει το κατάλογο μάλλον με την ελληνική κυβέρνηση. Έχουν πραγματοποιηθεί. Όσον αφορά τον κανονισμό στον οποίο είστε εισηγητής, Ζων ε, δεν πρόκειται να αναφερθώ. Αυτή η ιδέα να υπάρχει ένα νομικό σύστημα προστασίας τύπου, τύπου αν θέλετε, στο λεγόμενο Chapter 11, ε, κεφάλαιο 11. Νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να σας ενθαρρύνουμε να εργαστείτε προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, είναι καλό να μην τεθεί το θέμα ξανά, αλλά αν ξανατεθεί θα ήταν χρήσιμο να έχει στη διάθεσή μας ε, ένα προετοιμασμένο δρομολόγιο για να ξέρουμε ποια θα είναι η άουσα που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Λοιπόν, επί της αρχής συμφωνώ. Αλλά ξέρουμε και οι δυο και όλοι οι άλλοι ότι για την αρχή, επί της αρχής, είναι εύκολο να συμφωνήσουμε. Αλλά εγώ δεν είπα ότι δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα για την Ελλάδα. Γιατί αλλιώς θα δείτε στην που δεν σας αρέσει να βλέπετε. Uh, Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η Λίζα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βλέπω το, την παρουσία του κύριου Γιόγκρης εδώ πάλι και έχω δύο-τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, ελπίζω ότι το ESM θα ενισχυθεί Δεύτερον, αναφέρατε μακροοικονομικές ισορροπίες και ανισορροπίες. Πιστεύω ότι αν δούμε τον πίνακα ε, επιτυχιών, βαθμολόγησης δηλαδή, ε, εάν συμπεριφερθούμε έξυπνα, τότε θα επιτύχουμε ε, μια μεγάλη διαφορά. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά ως οικονομολόγος πιστεύω ότι το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα δεν μπορούσε να επιτύχει. Δεν είχε την ευκαιρία, το χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ σύντομο, ήταν υπερβολικά ακριβό και χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο για να εφαρμοστεί. Ε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να επιτύχει και έτσι οξύνθηκε η κατάσταση, οξύνθηκε το πρόβλημα. Τώρα ελπίζουμε ότι τα προβλήματα ε, έχουν περιοριστεί, ελέγχονται μάλλον και ότι περνάει μία φάση προσαρμογής ε, η όλη κατάσταση που στο τέλος θα επιτύχει. Βλέπουμε ότι δεν είναι δυνατόν λόγω της στασιμότητας που υπάρχει να επαναδιαπραγματευτούμε τις προθεσμίες που έχουμε αποφασίσει. Κάποιος πρέπει να μας πει, είτε είναι η Τρόικα είτε ο πρόεδρος του Eurogroup, ε, εσείς, ε, κάπως πρέπει να έχουμε τις απαντήσεις ενός νέου πακέτο που ελπίζω να οριστικοποιήθηκε τώρα πλέον. Δεν θα σας ζητήσω να μου πείτε ότι υπάρχει δυνατότητα τρίτου πακέτου, όμως θέλω να μου μου πείτε τι βιωσιμότητα και τι δυνατότητες υπάρχει στο δεύτερο πακέτο. Εάν το 2014 έχουμε ένα 2,5 πλεόνασμα, ε, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η βάση αυτής της προσδοκόμενης ανάπτυξης στην Ελλάδα, που θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του δεύτερου πακέτου. Επίση θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν ελάχιστε εγγύσεις για το PSI, που να μας δείχνουν ότι το PSI δεν θα μας οδηγήσει σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Διότι αν δείτε το πρόγραμμα, ρεαλιστικά δηλαδή, αυτό του οποίου έχει γίνει διαπραγμάτευση, θα πρέπει να ακούσουμε και τις απόψεις των πολιτών μας, τι χρειάζονται, τι θέλουν. Και πρέπει να έχουμε ένα σύστημα αντιμετώπισης ε, του χρέους μέσα στα πλαίσια της σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως με μία ατζέντα, με ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Ε, αν δείτε τις απόψεις που υπάρχουν στο κοινό, δηλαδή στο έδαφο, στη γη ας πούμε, στην πραγματικότητα, αυτά τα δύο στοιχεία δεν συμβαδίζουν, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η ελπίδα της ανάπτυξης και έτσι δεν, δεν υπάρχει και ε, εμπιστοσύνη στους πολίτες και αξιοπιστία. Δεν θέλω να απαντήσω στις λεπτομέρειες. Θα εξετάσω όμως υπάρχει κάποια μικρή διαφωνία όταν πρόκειται να εξετάσει η κατάσταση των ισορροπιών και των αντισορροπιών, όπως και εσείς και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε στις χώρες αυτές πιο ευρύ πρόγραμμα εξέτασης από ό,τι φαίνεται ότι διαφαίνεται αυτή τη στιγμή από τα κείμενα. Θα πρέπει να υπάρχει οριζόντιο ε, σε έλεγχο, ε, συγκρίνοντας τις χώρες, τις μεν με τις δε και δίνοντας κάποια στοιχεία ε, και τον και προς τα πίσω. Έχω πολύ κατανόηση για το γεγονός ότι ξεκινάμε από τη στιγμή κινήσης του ευρώ η κατάσταση ήταν διαφορετική κάποτε. Ακόμη και να εξετάσουμε το μοναδιαίο κόστος ε, των εργαζομένων, δεν αρκεί να πάρουμε σε σημείο κίνησης την 1η Ιανουαρίου 1999, θα πρέπει να ε, ανατρέξουμε μακρύτερα στο χρόνο. Γιατί η κατάσταση στις χώρες διαφέρει πάρα πολύ. Εγώ γνωρίζω κάποιες χώρες οι οποίες είχαν μία ανάπτυξη, αύξηση σημαντική του μοναδίου κόστους και συγκρίνεται με τους γερμανικούς ε, ε, παραμέτρους και υπάρχει ένα ε, νέο κόστος σε άλλες χώρες όπου αυξήθηκε με μεγαλύτερο ρυθμό ο μισθός από τη Γερμανία ε, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από την εκεί. Και βλέπουμε εκεί διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα από το που ξεκινάμε. Θέλω λοιπόν να υπάρχει συνεπής ε, εξέταση. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι παρουσιάζοντας τις εκθέσεις αυτές θέλει κανένας να πιέσει τους εξεταστές προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και γι' αυτό πρέπει κανένας να αναρωτηθεί όσον αφορά την μέθοδο που χρησιμοποιείται. Θεωρώ ότι στο δεύτερο πρόγραμμα για την Ελλάδα οι διαστατικές ε, μεταρρυθμίσεις είναι πολύ πιο σημαντικές από ότι στο πρώτο. Εν τω μεταξύ υπάρχει βέβαια ο χρόνος που έχει οδήγησε κάποια αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν πολλά διορθωτικά προγράμματα που έχουν απαριθμιστεί στις ε, πράξεις ε, προτεραιότητας που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη ανάπτυξη. Βέβαια, με μονομένα τα διορθωτικά προγράμματα προχωρούν προς την καλή κατεύθυνση, θα πρέπει να εξετάσουμε όμως το σύνολο. Είδατε ότι η, ε, το Eurogroup αναφέρεται σε κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, αποφάσεις που πήρε μέσα στα πλαίσια του πρώτου προγράμματος. Ε, μειώθηκε το επιτόκιο που εφαρμόζεται για την περίοδο 2012-2020 μειώσαμε τα επιτόκια που είχαν αρχικά οριστεί για να δοθούν περισσότερες δυνατότητες εξυγένσης στην Ελλάδα στα 8 πρώτα χρόνια του προγράμματος παγίωσης. Για την ανάπτυξη δεν σας είπα ό, όλο αυτό που σας να πει, εξέφρασα την άποψή μου, γιατί σας είπα ότι δεν πρέπει να γίνει κριτική, αλλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε προτάσεις. Για τα ευρωομόλογα είπα λίγο πολύ ότι είχα να πω. Υπάρχουν εκεί πιο άμεσα αποτελέσματα με μια αυθόρμητη απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από την Άλντι Σιλβή. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε στην Καθολική Εκκλησία, διότι επιτέλους κατάλαβα ποια, ποιο είναι τα σημεία αναφορά σας και κατάλαβα γιατί το Συμβούλιο των, ε, των Διοικητών της Κεντρικής Τράπεζας αποτελείται μόνο από Έλληνες. Ήμουν από τα μέλη του Κοινοβουλίου που εκφράσαμε την επιθυμία μας όταν μας παρουσιάζεται ε, υποψηφίους για το Συμβούλιο να έχουν περισσότερες γυναίκες. Τώρα, σχετικά με την Ιρλανδία. Ε, κοιτάξτε, εγώ σέβομαι τις αποφάσεις όλων, αλλά ε, θα πρέπει να σκεφτούμε συλλογικά και ανησυχώ πολύ με αυτά που είπατε κύριε Πρόεδρε. Ανησυχώ πράγματι, διότι είχαμε ήδη την, την εμπειρία αυτής της προσπάθειας ε, των στεγανών σε ό,τι αφορά την ε, Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με συνθήκες που αφορούν όλους τους πολίτες των χωρών να ρωτάμε τη γνώμη των μεν και όχι των δε και αν έχουμε χωριστές ε, διαδικασίες ε, πιστεύετε ότι θα προχωρήσουμε θεωρείτε ότι βρισκόμαστε στο πλαίσιο δημοκρατικών αρχών που για ένα θέμα κοινού να υπάρχει ε, ένας άνδρας, μια γυναίκα, μια ψήφος και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πολύ καλά τα εθνικά συντάγματα. Καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά συνεχίσουμε ότι ούτω τρόπος θα διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα μια χώρα που ε, εφάρμοσε τα δημοσφίσματα. Δεν θέλω να δώσω μάθημα σε κανέναν. Απλά λέω ότι είναι μια αντίληψη της δημοκρατίας που δεν ε, ταιριάζει με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και που θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στις αγορές. Ο κ. Ντράγκη το είπε εδώ, ότι έχουμε ανάγκη από ένα fiscal compact, ένα σύμφωνο δημοσιονομικό. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω πως ε, παρά τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουμε τη στιγμή, συμμετοχή γυναικών στο Συμβούλιο θα, αποτε... θα αποτελέσει πολύ λιγότερη προσπάθεια από ότι η συμμετοχή γυναικών στην Καθολική Εκκλησία. Μιλάω για τον κλήρο. Τώρα, σε ό,τι φορά την ε, Ιρλανδία, Σιλβί, μια που καθημερινά σχεδόν ε, διαβάζω τα άρθρα σας ε, που είναι εξάλλου υψηλή ποιότητα, ότι οι χρηματαγορέ θα πρέπει να σέβονται τη δημοκρατία. Εγώ έχω βαρεθεί να το επαναλαμβάνω, πως ε, σε κάθε στιγμή θα πρέπει να διερωτώμεθα για το πώ αντιδρούν οι χρηματαγορές. Η δημοκρατία ζει, κινείται. Και δεν μπορούμε κάθε φορά να μια Μα αυτές καθημερινά με ταράζουν. Αλλά εσείς θίξατε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δηλαδή η προσφυγή σε ένα δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ταραξει τις αγορας μα αυτες καθημερινα μεταράζουν. αλλα εσεις θιξατε ενα υπαρκτο προβλημα δηλαδη η προσφυγη σε ενα δημοψηφισμα δεν ειναι κατι το οποιο μπορει να σταθεροποιησει στο σύνολο την, σύνολο, την πολιτική κατάσταση στη ζώνη ευρώ. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτή τη φορά το Ιρλανδικό δημοψήφισμα δεν θα προκαλέσει τις ίδιες ε, τραγικές ε, επιπτώσεις ε, που είχαμε με προηγούμενα δημοψηφίσματα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Το ζήτημα είναι υπαρκτό, αλλά δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσουμε. Και εγώ το βλέπω με τον ίδιο τρόπο που και εσείς, αλλά δεν θα πρέπει να κλείνουμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ένα δημοψήφισμα σε κάθε κράτο μέλο κάθε φορά που θα επανεξετάζουμε τι ε, συνθήκε. Το 2005 μετά από το ε, γαλλικό και ολλανδικό όχι, γνωρίζω όλες τις ε, διαδικασίες που μπορεί να φαίνονται αρχικά απλές, αλλά τη απουσία μιας συνθήκης μπορούν να περιπλακούν επικινδύνως όταν ένα κείμενο επιβάλλεται στην αξιολόγηση των ε, πολιτών. Ε, όμως ε, ένα δημοσιονομικό σύμφωνο δεν περιλαμβάνει ψηλό αριθμό άρθρων και σε ό,τι φορά το περιεχόμενο έχει αναφορές στο παράγωγο δίκαιο που ήδη υπάρχουν. Άρα λοιπόν η όλη προσπάθεια θα μπορεί να συνοψιστεί σε πολύ λίγα. Ευχαριστώ. Ο Σβέν. Α. Κυρία Πρόεδρε, με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τα σχόλια για την Καθολική Εκκλησία. Εγώ είμαι καλβινιστής και με αυτή τη βάση θα συνεχίσω. Εγώ νομίζω ο κύριος Γιούγκερ έχει γίνει Ευρωπαίος Πάπας, ε, κάπως έτσι. Βρίσκεται παντού και πουθενά. Παντού. Ο κύριος Ολόντ που είναι υποψήφιος των σοσιαλιστών είπε ότι θέλει να επαναδιαπραγματευτεί αυτό το δεύτερο πακέτο όσο έχει συμφωνηθεί και χτες έγινε μια συζήτηση και ακούστηκαν πολλές επικρίσεις από την αριστερά, από τους σοσιαλιστές, τους Γάλλους σοσιαλιστές, ε, τους πράσινους, ε, τις μη τα μη ορθόδοξα αριστερά κόμματα τα οποία είναι υπέρ του ευρώ αλλά κατά των επιπτώσεων του ευρώ. Αυτό ας το σκεφτόντουσαν πριν από δέκα χρόνια η νομισματική ένωση χωρίς ένωση των προϋπολογισμών δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει και γι' αυτό ακριβώς κάναμε και την εισαγωγή αυτού του δημοσιονομικού πακέτου. Ως κάποιος ο οποίος έχει ζήσει κάποτε σε μια χώρα που υπήρχε ένα τσάρο. Ο κύριο Σολόντι είπε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, αλλά υπάρχει εναλλακτική λύση. Έτσι δεν είναι sans Δίχως να θέλω να έχω μια κάθετη αντιμετώπιση, θα σας πω ότι ως χριστιανοδημοκράτης δεν θεωρώ πως περιγράφεται την θέση των Γάλλων Σοσιαλιστών με σαφή τρόπο και ακριβή τρόπο. Πάντως ε, ε, σας ε, συγχωρώ, όπως και σε όλους τους αμαρτωλούς. Δεν γνωρίζω τα, ακριβώς ε, τα, τα του κυρίου Ολόντ, αλλά παίρνω σοβαρά αυτά που λέει. Και με αναζωογονεί, διότι το 97 ο κύριος Σιράκ ε, σε μια δύναμη θέση ε, προέβη στην διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και άνοιξε τις πόρτες ε, της Πρωθυπουργίας στον κύριο Ζωσπάν και σοσιαλιστές και είχε πει τέτοια πράγματα με αυτά που λέει ο κύριος Σολών για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Το Λουξεμβούργο τότε είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω λοιπόν πώς μπορούμε να απαντήσουμε στις ε, επιθυμίες ε, του Γαλλικού Συντηρητικού Κόμματος και θα πράξουμε το αυτό. Εάν ε, συμβεί κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, για το οποίο δεν είμαι και πολύ φανατικός υποστηρικτής, δεν μπορεί να τύχει επαναδιαπραγμάτευση στο σύνολό του. Είναι προφανές πως μια αναπτυξιακή πολιτική δεν ε, διατάσσεται μέσω άρθρων, δεν μπορείτε με συνθήκες, δεν μπορείτε μέσω ενός άρθρου να καθορίσετε την αναπτυξιακή πολιτική, ενώ είναι πιο εύκολο να έχετε μια δημοσιονομική πολιτική μέσω συγκεκριμένων διατάξεων μιας συνθήκης. Θα δούμε λοιπόν όταν φτάσει η στιγμή. Είχαμε μια κατάσταση αντιμετωπίσει το 1997 και θα ζητήσω στον καλβινιστή φίλο μου να παραμείνει πιστός. Να μην απαρνηθεί την πίστη του. Τώρα Σβέν. Ζαν κλοντ Juncker, η εντύπωση μου είναι ότι το Συμβούλιο και το Ευρωγκρουπ συγκεκριμένα έχουν παρερμηνεύσει την ελευθερία του χριστιανού ανθρώπου. Διότι η κεντρική ιδέα είναι ότι τα, τα πάντα δικαιολογούνται λόγω της πίστης και όχι από τις πράξεις. Αυτή ήταν τότε η μεγάλη επανάσταση της μεταρρύθμισης. Τώρα ας δούμε το μόλις μεταρρυθμισμένο σύμφωνο ε, σταθερότητας. Έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζονται αυτοί οι κανονισμοί. Στην Ισπανία είχαμε 8,5 έλλειμμα για το 2011 και Τώρα ε, του χρόνου θα είναι 8,4 το έλλειμμα αυτό και η Ισπανική κυβέρνηση λέει ενώ ο στόχος ήταν η μείωση σε 6% δεν μπορεί να το επιτύχει τώρα. Στην Πορτογαλία πέρσι είχαμε στόχο 5,9%, κατάφεραν 4% αλλά μόνο 3,5% τελικά ε, πραγματοποιήθηκαν με τα μέτρα που εφάρμοσαν. Πέρσι ελπίζω να τα καταφέρουν φέτος. Τώρα σας ρωτώ, εσείς συνεχίζετε και πιστεύετε και έχετε τις ελπίδες σας μόνο στην πίστη ή πιστεύετε ότι, ελπίζω να μην πιστεύετε, το πρόγραμμα αυτό το, μεταρρυθμιστικό να καταλήξει να, είναι μια σκιά μόνο ε, στο μέλλον. Πώς θέλετε να συγκεράσετε την πραγματικότητα με τη, θεωρία, την πράξη με τη θεωρία, δεδομένου ότι τα ελλείμματα βλέπουμε ότι αυξάνονται, αντί να μειώνονται. Πότε επιτέλους θα συμβαδίσουν τα μέτρα δημοσιονομικού περιορισμού, με μέτρα ανάπτυξης, με μέτρα ενίσχυσης, ε, μέτρα δηλαδή τα οποία θα δώσουν ε, ουσία, θα δώσουν κόκαλα αν θέλετε στο σύμφωνο σταθερότητος. Ο κύριος Γιόγκερς. μέχρι σήμερα, πριν από λίγα λεπτά, Α, δεν ήξερα ότι εδώ η επιτροπή ευτύπου που και που γίνεται και θεολογικό, μετατρέπεται μάλλον σε θεολογικό σεμινάριο. Ο Θεός, ο Θεός να έχει καλά την Ευρώπη δηλαδή. Πάντοτε ήταν δυνατή η πίστη στην Ευρώπη. Και με την ελπίδα και μόνο δεν θα πετύχουμε. Ελπίδα και αγάπη, ομόνοι, όλα αυτά δεν φτάνουν. Εντάξει, γιατί όχι μόνο πίστη, αλλά και αγάπη. Ε, η αγάπη όλο και μικραίνει στην Ευρώπη, περιορίζεται, όλο και λιγότερο αγαπιόμαστε. Και ποτέ δεν πίστευα ότι στην Ευρώπη θα ήταν δυνατόν ακόμα Να υπάρχει έξτρα, τέτοια έξτρα έναντι ορισμένων κρατών μελών. Περισσότερη αγάπη λοιπόν χρειαζόμαστε. Για, όσον αφορά την Ισπανία, ε, έχουμε μία ε, ξεκάθαρη εικόνα και αύριο θα κάνουμε μία δήλωση, ε, θα ακούσουμε τη δήλωση του Ισπανού Υπουργού Οικονομικών και μέσα στο σύμφωνο σταθερότητος ισχύει και το εξής. Στην αξιολόγηση του ελλείμματος δεν πρέπει να αγνοούμε όλους ε, τους συναφείς παράγοντες Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφείς εξηγήσει, να ξέρουμε ποιοι παράγοντες οδήγησαν στο να εμποδίσουν την Ισπανία να τηρήσει το στόχο της για το 2011 και να μην μπορέσει να μειώσει, να φτάσει δηλαδή τα ποσοστά που ήθελε. Ε, Α μην ε, ξεχνάμε και την πλευρά του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Ε, το οποίο ισχύει βεβαίως στην Ισπανία σφαιρικά, πέραν των προβλημάτων που έχει στις ε, περιφέρειες και στις αυτόνομες περιοχές, πρέπει για την Ισπανία να δούμε πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον οι υπολογισμοί και τα οικονομικά αναπεριφέρεια. Ε, εγώ δεν είμαι σεσμός ούτε φορές είναι, είμαι απλώς ένας μικρός δευτερεύων Άγιος σε μια Αγία μεγάλη οικογένεια. Οπότε ε, έχω και έναν περιορισμένο ας πούμε ρόλο. Δεν νομίζω όμως ότι τα προβλήματα στην Ισπανία είναι τόσο αξία όσο παρουσιάζονται και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός εχθές, ο Υπουργός Οικονομικών, συγγνώμη, δήλωσε ότι δεν επισημεί η Πορτογαλία να ζητήσει την επιβολή επιπλέον προγραμμάτων ή την παροχή επιπλέον προγραμμάτων. Δεν θα ζητήσει επιπλέον μέτρα και προγράμματα. Δεν πιστεύω ότι ε, μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε μία ομόνια μεταξύ μας. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ε, δεν αρέσει, αλλά πρέπει να πω ότι ορισμένες ιδέες δεν είναι επικοδομητικές. Ε, αυτές που άκουσα τις τους τελευταίους 14 μήνες ελπίζω να διαψευθούν οι κακοί ιονοί ε, και να διψευθούν όλοι αυτοί που θέλουν να επιβεβαιωθούν οι δυσμενείς προβλέψεις τους. Δεν είναι παρηγορία, αλλά κάτι είναι και αυτό. Πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας, λέει η Πρόεδρος. Τώρα για την ΚΟΕ ο κύριος Χουντής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ, σε συνέντευξή σας σε γερμανική εφημερίδα δηλώσατε αν στην Ελλάδα ενισχυθούν ακραία κόμματα σε βαθμό που το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να φτιάξουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αυτοί που θα κυβερνήσουν θελήσουν να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα σωτηρίας θα αποχωρήσει και η Ευρώπη και σε άλλη συνέντευξη συμπληρώσατε ότι χρειάζεται να υπάρξει επίτροπος για την Ελλάδα θέλω να σας πω ότι ο εκβιασμός σας είναι για τους Έλληνες προφανής τι μας λέτε. Πρώτον, ή ψηφίζετε τα κόμματα που στηρίζουν σήμερα το μνημόνιο και που δεν είχαν το θάρρος, δεν είχαν την αντοχή να υπερασπιστούν τον ελληνικό λαό από την ταπείνωση ή τώρα που εξασφαλίσαμε τις τράπεζες, τώρα που εξασφαλίσαμε την επικυριαρχία με επιτρόπους και γκαουλάιτερ, τώρα που σας έχουμε σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας, να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε την κυβέρνηση και το κόμμα που σας ανήκει. Δηλαδή, μας υπόσχεστε επιλεκτική δημοκρατία. Και πού το λέτε αυτό, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Πριν λίγους μήνες θα έλεγα στον πρόεδρο της Ευρωζώνης ότι η θέση του δεν του επιτρέπει να κάνει τέτοιες αγενείς δηλώσεις. Θα του έλεγα ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να χαρακτηρίζει ακραίο κάθε άλλο ελληνικό κόμμα εκτός από το Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία θα του έλεγα ότι δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να μας επιβάλλει ποια κυβέρνηση θα έχουμε στην Ελλάδα. Δεν σας τα λέω αυτά, όχι γιατί δεν γνωρίζω το βαθμό αγιοσύνη σας και κάνετε χιούμορ με αυτό, αλλά γιατί αναγνωρίζω στο πρόσωπό σας έναν άξιο εκπρόσωπο μιας Ευρώπης που έχει διαμορφώσει ένα τραπεζικό και δημοσιονομικό νταχάου, έναν κοινωνικό και εργασιακό μεσαίωνα, μιας Ευρώπης της ιδεραίας πειθαρχία μιας γερμανικής Ευρώπης. Γι' αυτό αγαπητέ κύριε Γιούγκερ δεν σας ρωτάω από πού αντλείτε αυτό το δικαίωμα να κάνετε αυτές τις αγενείς δηλώσεις για την πατρίδα μου. Euh, Μ' αρέσει να απαντώ με τρόπο απλό στις περίπλοκες απαντήσεις αλλά και το αντίστροφο. Εάν ε, αυτό σας βολεύει να παρουσιάζετε τα λόγια μου με τον τρόπο που το πράξατε και αυτό θα πρέπει να σας βολεύει διότι δεν υποτιμώ την ε, ικανότητα ερμηνείας ε, ενός ε, κειμένου που σας υποβλήθηκε. Τότε δεν έχω καμία τύχη να σας εξηγήσω, για να σας εξηγήσω λεπτομεριακά τι δήλωσα σε μία γερμανική εφημερίδα, τη συζήτησα με τα κόμματα του κυβερνητικού συντασπισμού και τι είπα σχετικά με τα ζητήματα που θίξατε. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω εξτρατεία για τα δύο κυβερνητικά κόμματα, διότι κρίνω ότι και τα δύο είναι απολύτω υπεύθυνα για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Δεν έχω κανένα λόγο να επικρατώ του σοσιαλιστέ και του Έλληνε συντηρητικού, γιατί θα το πράταξα το Λεχθάντος, ε, τα δύο αυτά κόμματα ε, συναποτελούν ε, τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ζήτησα την υπογραφή του κυρίου Πανδρέου και του κυρίου Σαμαρά, τον οποίο συναντήσω και αύριο το πρωί και δεν μπορούσα, πώς να το πω, να τρέξω πίσω από όλες ε, τις ε, πολιτικές ε, θέσεις της Ελλάδας. Εσείς εκπροσωπείτε την πλέον έντιμη, την πιο άξια ενδεχομένω άποψη. Μπορούν να λένε οι ε, τα κόμματα τα οποία θα είναι στην κυβέρνηση ότι δεν δέχονται το πρόγραμμα, εντάξει, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, υπάρχει όμως δημοκρατία και στις υπόλοιπε 16 χώρες της ζώνης ευρώ. Και μία δημοκρατία δεν αξίζει περισσότερο από την άλλη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ευαίσθητοι στις αντιδράσεις συνάψαμε μια συμφωνία και ένα πρόγραμμα με την ελληνική κυβέρνηση στη δημοκρατία αλλά και σε άλλα καθεστώτα υπάρχει ο κανόνας της συνέχισης του δημοσίου και το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί από η ελληνική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις ε, εκλογές ε, του ε, Απριλίου ή αργότερα. Εγώ δεν συμφώνησα με την αποστολή ενός ε, επιτρόπου στην Ελλάδα. Ε, επίτροπο εξοικονόμησης τώρα, να διορίσουμε τώρα έναν επίτροπο στην Επιτροπή, στην Κομισιόν, που θα ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με την ε, πολιτική προώθησης, ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τα προβλήματα είναι τέτοια φύσης και η απελπισία, η απόγνωση του ελληνικού λαού είναι πολύ σοβαρή και θα μπορούσε να αναλάβει ένας ε, επίτροπος ε, το θέμα της ανάπτυξης και να αποκτήσει όλες τις ε, αρμοδιότητες προκειμένου μια ουσιαστική στρατηγική προσδεύση αυτή να εφαρμοστεί. Λοιπόν, μη συγχαίρεται επίτροπο με επίτροπο, μη συγχαίρεται με αυτό το οποίο πρότεινα και επαναλαμβάνω, αν το να πούμε ότι παράλληλα με τις πολιτικές ε, στήριξης ε, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός και διοικητικός μηχανισμός ο οποίος ε, θα φροντίσει ώστε οι πολιτικές ανάπτυξης να μην παραμείνουν στο στάδιο των επιθυμιών, αλλά να υπάρξει πρόοδος και που θα ξαναδώσει ελπίδα στους Έλληνες πολίτες. Δεν είμαι πρόεδρος στην Κομισιόν, ο κ. Μπαρόζο είναι, σε αυτόν το είχα πει, δεν μπορώ να επηρεάσω τα πράγματα, απλά εγώ προτείνω. Αυτό είναι το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος από το EFD θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Γιούγκερς που είσαστε εδώ κοντά μας σήμερα. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι σκέψεις για τη σημερινά γεγονότα. Πριν από λίγες ώρες πριν έρθω εδώ, διάβασα στο διαδίκτυο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, προβλέπει πάλι, έδωσε μάλλον, έριξε 500 δισεκατομμύρια ευρώ στις αγορές Αυτό σας ανησυχεί, σας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις όσον αφορά τον πληθωρισμό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει όσο πάει και περισσότερο την ιδέα του έσχα του ε, δανειστή για τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Απάντηση. Ποτέ δεν προτίθεμαι να σχολιάσω αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρική Τράπεζα. Το ξέρετε. Ακόμα και αν πολλές φορές συμφωνώ απόλυτα με την έκτα, δεν θα έλεγα ότι αν έπρεπε να εκφραστώ επ' αυτού θα ήταν αυτή η περίπτωση, αν ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεύτερο, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορέσει να αποσύρει από το ε, κύκλωμα αυτά τα ποσά που οδηγούν πραγματικά σε πληθωρισμό. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Για τις επόμενες ερωτήσεις θα πρέπει να τις συνενώσω νομίζω και παρακαλώ όλους να μην μακρηγορήσουν και εσείς Jean-Claude μετά παρακαλώ. Τρεις ερωτήσεις Παρότι τα και ο Μπούλμαν. Ο Παύλο πρώτα. Σε ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ, θα αναφερθώ στην Ισπανική στην χώρα μου, την Ισπανία. Η Ισπανία σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έκανε τρεις μεταρρυθμίσεις σημαντικές. Σταθερότητα στον προπολογισμό, ε, ε, μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματο και εργατική μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω, Πρόεδρε Γιούνκερ, την αξιολόγηση από πλευρά σα. Εξάλλου όλοι συμφωνούμε πω μόνο με λιτότητα, μόνο με περικοπέ, μόνο με κλείσιμο των χασμάτων των τρυπών δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Εσείς για μια πολιτική ανάπτυξη για την Ελλάδα. Ε, Εμεί συμφωνούμε ότι όχι μόνο είναι απαραίτητη για την Ελλάδα αυτή η πολιτική, αλλά και για την Ισπανία. Υπάρχει ένα, μια επιστολή την οποία γνωρίζετε 12 πρωθυπουργών μεταξύ αυτών και το δικού μου ζητώντας από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να δώσει έμφαση στο ζήτημα της ανάπτυξης. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ, και εγώ θα ήθελα να... Θα ήθελα να σας πω πόσο σου αρέσει να σας ακούω όταν ερχόσαστε εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να περάσω πάλι στο θέμα της Ιρλανδίας και το θέμα του διποψηφίσματος. Γιατί αναφερθήκα σε δύο σημαντικά θέματα, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα του δημοψηφίσματος και ο συσχετισμός ε, του δημοσιοποιήσουμε την πρόσβαση της, ε, της Ιρλανδίας στο Ταμείο Σταθερότητας. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως. Οι επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο αρνητικό δημοψήφισμα στην Ιρλανδία θα έχει στη δυνατότητα στο μέλλον να ενταχθεί η χρηματοπιστωτική ε, δημοσιονομική συνθήκη στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εάν υπάρχει αρνητικό δημοψήφισμα δεν θα μπορεί αυτή η συνθήκη να ενταχθεί στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό με κάνει να περάσω στη δεύτερη μου ερώτηση. Ποιο, τι πιστεύετε για τον ενδεχόμενο κίνδυνο στο μέλλον να υπάρχει πιο συχνά πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο της διακυβερνητικής συμφωνίας Ευχαριστώ, Ουντο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Γιούγκερ, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του Επιτρόπου Ανάπτυξης. Εγώ το κατάλαβα διαφορετικό το θέμα από ότι ο Έλληνας ε, συνάδελφος που μίλησε. Γιατί εάν προχωρήσουμε με τη σκέψη αυτή που θέλω να κάνω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι θετικό, μια ευκαιρία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν, όσον αφορά την ιδέα της ε, ε, βοήθειας για την Ελλάδα, θα πρέπει να βγούμε από μια, ένα σκεπτικό σύμφωνο με το οποίο αμέσως υπάρχει ε, το αποτέλεσμα των επιδοτήσεων και η ανάπτυξη αργότερα, μήπως θα πρέπει να υπάρχει μια ε, διεύρυνση της δικής σας πρότασης αν αυτός ο νέος επίτροπος ε, υποβάλλει αυτό το νέο σημείο για συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αυτό θα κλείσει και ένα δημοκρατικό κενό που υπάρχει. Μερικέ απαντήσει παρακαλώ. Όσον αφορά την ερώτηση του Παύλου και τι ε, που είχε η Ισπανία τους τελευταίου μήνες, εγώ γενικά ομολογώ ότι είμαι ικανοποιημένο από τι πολιτικέ αποφάσει που ελήφθησαν στην Ισπανία. γιατί κατευθύνονται προς την κατεύθυνση της παγίωσης, αποδεικνύουν ότι η Ισπανική κυβέρνηση είναι σταθερά αποφασισμένο να εγκαθιδρύσει μια πολιτική παγίωσης και γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να επικρίνουμε την κυβέρνηση κ. Τραχώη για την πολιτική αυτή που ακολουθεί. Δεν μπορώ να διαβάσω εδώ τι έχω σημειώσει για τη δεύτερη σας ερώτηση. Για πέστε μου τι ήταν η δεύτερη σας ερώτηση. Για... Την αξιολόγησή σας, την άποψή σας σχετικά με την επιστολή που έστειλαν ορισμένοι πρωθυπουργοί. Α, ναι, ναι, ναι. Είχα σημειώσει μόνο το 12 και δεν ήξερα τι ήταν αυτό το 12. Ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική ο αριθμό σα. Εγώ δεν υπόγραψα αυτή την επιστολή. γιατί λείπουν κάποιες απλές λέξεις. Ε, κοινωνική διάθεση, στάση, παραδείγματος χάρη. Εμένα με τρόμαξε αυτή η έλλειψη της κοινωνικής διάστασης σε αυτό το κείμενο. Η Ντανούτα μου υποβάλλει κάποιες ερωτήσεις ουσιαστικότατες. Ας πούμε, ότι δηλαδή θα πει όχι στο δημοψήφισμα. Αυτό τι θα σημαίνει. Ότι δεν θα μπορούμε πια να εισαγάγουμε τις διατάξεις της διακυβερνήσεως αυτής στην βασική σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν θα ήθελα να το κάνουμε. Το είπα πολλές φορές. Εμένα δεν μ' αρέσει η διακυβερνητική προσέγγιση. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε μια κοινοτική προσέγγιση ειλικρινά. Αλλά ακόμα και αν η Ιρλανδία πει όχι, το θέμα θα ξανατεθεί στον Ιρλανδικό λαό όταν προσπαθήσουν να εισαγάγουν τις διατάξεις αυτές στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι εάν την πρώτη φορά πει όχι ολό θα πρέπει να ξανααποφασίσει και το έχουν ξανακάνει και στο παρελθόν. Α, τώρα, αυτός ο, ο Επίτροπος Ανάπτυξης, όπως είπατε, θα έπρεπε, έτσι το είχα σκεφτεί τουλάχιστον, να είναι ένας ε, θετικός παράγοντας όχι κάποιος τιμωρός που θα αποσταλεί στην Ελλάδα, αλλά κάποιος που θα είναι ο φίλος των Ελλήνων και θα τους ε, βοηθήσει να ξαναβρούν ε, στοιχεία ανάπτυξης. Και πιστεύω ότι εάν υπήρχε ένας τέτοιος επίτροφος, οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου για την εξέταση της στρατηγικής αυτής. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο Επίτροπος Ανάπτυξης ακόμα και ακόμα και αν υπήρχε δεν πρόκειται εγώ να του πω τι θα κάνει. Αλλά αν έχει νόημα αυτό το καθεστώς θα πρέπει πραγματικά να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα είπαμε. Πρόεδρος, ωραία. Δύο ενότητες, δύο ερωτήσεων. Η Άστρη Λουλίν και μετά η Άννη Ποδηματά. Πρώτα η Άστρετ. Κύριε Γιούνκερ, σε ό,τι φορά την πρόταση να διορίζει ο κ. Μπαρόζο έναν επίτροπο που με την ανάπτυξη της Ελλάδας, ίσως ε, να σας υπενθυμίσει αυτό που ο Βίκτορ Ουγκό είχε πει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από μία ιδέα την κατάλληλη στιγμή. Ίσως αυτή η στιγμή να έχει φτάσει. Μέσα τόσο στην περίπτωση της Ελλάδας και την ενδεχόμενη επιτυχία στο έργο αυτού του Επιτρόπου να υπενθυμίσω πως οι εμπειρίες του παρελθόντος μας κατέδειξαν ότι οι διασώσεις των χωρών που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν εστέφθησαν από επιτυχία παρά μόνο ε, τα μέτρα μείωσης των δαπανών συνοδεύονται από μια ε, νομισματική υποτίμηση. Και στο πλαίσιο του ενιαίου νομίσματος αυτό είναι είναι δυνατόν, ενώ, εκτός αν η Ελλάδα βρει βγει από το ευρώ, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό για πολλούς λόγους, τους οποίους και στηρίζω. Αν δεν υπάρχει λοιπόν υποτίμηση, πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε μια βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, διότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κανένα παράδειγμα στην Ιβίλιο εκτός αν πιστεύουμε στα θαύματα. Πώς βλέπετε πρόεδρε τα πράγματα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε τα πράγματα να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση ενώ οι κακές ειδήσει αποθαρρύνουν και τους πλέον αισιόδοξου. Ανή. Ευχαριστώ Πρόεδρε να σε ευχαριστήσω για τις ε, πληροφορίες και για τις αποφάσεις που λάβατε σχετικά με την Ελλάδα. Ιδιαίτερα διότι τονίσατε πως η Ελλάδα χρειάζεται μια αναπτυξιακή πολιτική προκειμένου να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις ε, των δημοσιονομικών περικοπών ε, Α, θέσω ένα ερώτημα. Όχι, δεν θα θέσω ερώτημα σχετικά με το κόμμα, διότι γνωρίζετε πολύ καλά τα πράγματα. Τα κόμματα στην Ελλάδα, αναφέρατε το Πασόκη η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτά τα οποία φέρουν την ε, ευθύνη της κατάστασης. Συμφωνώ μαζί σας, χωρίς να αποκλείω φυσικά και της, τη συμμετοχή και των κομμάτων της αριστεράς στην κατάσταση αυτή. Να θέσω ένα ερώτημα λοιπόν εξ ονόματος των Ελλήνων πολιτών τουλάχιστον εξ ονόματος εκείνων που είναι υπέρ της Ευρωζώνης και της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη όπως το καταδεικνύουν και οι πρόσφαρες να σας ζητήσω να τους απευθύνετε ένα μήνυμα, διότι αυτοί, όπως είπατε, πολύ σωστά φέρουν το βάρος σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της χώρας. Διότι κανένα πρόγραμμα ή ε, καμία δημοσιονομική λιτότητα, καμία στρατηγική δεν να πετύχει χωρίς, μάλλον αν συνεχίσουμε αυτή, αυτές τις ε, συζητήσεις ανταλλαγής ε, επιχειρημάτων, θα τα καταφέρει η Ελλάδα, θα τα καταφέρει, θα χρεοκοπίζει ή όχι θα ενθαρρυνθεί ή θα της επιβληθεί η έξοδος από το ευρώ. Εάν συνεχιστεί λοιπόν αυτή η κατάσταση, δεν υπάρχει καμία επιτυχία να πετύχει το οποιοδήποτε πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Να πω στην Άστριντ ότι ο Βίκτορ Ουγκό έγραψε την πρόταση που ανέφερες στην στην εξορία του όταν βρισκόταν στο Λουξεμβούργο. Εμπνεόταν ο Βίκτορ Ιγκό όταν εκδιώκεται από την Γαλλία, όταν εγκατέλειπε τη Γαλλία. Εκτός μικροφώνου κυρία Λούλινγκ. Δεν ήταν στο Λουξεμβούργο. Αν επισκεφθεί στο Λουξεμβούργο <laughs> και αν μείνει πάνω από τρει μέρε, θα έχει επισκεφθεί όλε τι πόλει και όλα τα χωριά του. Τουλάχιστον ο Ούγκο γνώριζε που ήταν το Σέγγεν, διότι μια μέρα ο Μητερό στην γαλλική τηλεόραση είπε ο, κανείς δεν ξέρει τι είναι το Σέγγεν, βρίσκεται στις καντοχώρες, κάτι το οποίο έκανε λάθος, αρκεί να διάβαζε που βρισκόταν ο Βίκτορ Ιγκό συχνά. Τα είχε μάθει περισσότερα για την γεωγραφία του Λουξεμβούργου. Τώρα η περίπτωση της Ελλάδας είναι μοναδική ε, έκτακτη, διότι ποτέ δεν είχε υπάρξει νομισματική ένωση του είδους της δικής μας και δεν υπήρξε μια χώρα που διολίστησε αλλά η Ελλάδα έχει προβεί σε μια εσωτερική υποτίμηση. Και να επαναλάβω ότι φυσικά θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ και μια πραγματική προσπάθεια ανάπτυξης. Ε, το λέμε εύκολα, αλλά δεν είναι, γίνεται στην πράξη εύκολα. Γίνεται δύσκολα στην φάση, διότι η δομή της Ελλάδας ε, δεν, παρο... δεν μοιάζει με τη δομή των οικονομίων των άλλων κρατών μελών της ζώνης ευρώ. Είναι πολύ αδύναμη η προσπάθεια λοιπόν που θα πρέπει να καταβληθεί, θα πρέπει να είναι έντονη και εντατική. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα τον ορισμό ενός επιτρόπου που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα που είναι τόσο σημαντικό για τους Έλληνες αλλά και για μας. Η Ιρλανδία πράττει σωστά. Θα ήθελα και η Ελλάδα να κάνει το ίδιο. Απάντω και Ζωχάνες. Εάν η Ιρλανδία αποδεικνύει πως ε, κατορθώνει να αντιστρέψει την κατάσταση. Φυσικά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιρλανδία και οι αιτίες είναι εντελώς διαφορετικές. Θα πρέπει όμως ε, ο, μαζί να προσπαθήσουμε η Ελλάδα να αποτελέσει ένα παράδειγμα η οποία θα αποδείξει όταν φτάσει η ώρα ότι οι προσπάθειες δεν ήταν μάτιες, ούτε οι προσπάθειες των Ελλήνων, ούτε οι δικές μας. Και εντάξει, συμφωνώ απόλυτα θα πρέπει να σταματήσουμε αυτήν την πολυλογία για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας ε, από τη ζώνη ευρώ. Εξάλλου όσοι το κάνουν αυτό, δεν το κάνουν με βάση μια ανάλυση σε βάθος, αλλά για λόγους εκλογικούς ε, που αναφέρονται στον ορίζοντα. Έχουμε μια νομισματική ένωση με 17 μέλη. Η έξοδος της Ελλάδας δεν είναι μια υπόθεση εργασίας. Εάν δεν ήταν τόσο οδυνηρό, θα σας έλεγα ότι ε, ο καθολικισμός λέει ότι υπάρχουν ερωτήματα που δεν τίθονται. Αλλά δεν θα ήθελα να κάνω, σας κάνω μια υπερβολική δόση ε, καθολικισμού στην συνεδρία. σας. ευχαριστώ πολύ. Σύντομες ερωτήσεις, Λάμπερτ και Γκουαλτιέρη. Σύντομα παρακαλώ, διότι ο Ζων Κλοντ έχει ακόμα μισή σελίδα από το σημείο το, το ξενοδοχείο Σοφιτέλ. Ε, τώρα, εάν ε, πάμε στην Ελλάδα και πούμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι μισθοί, η Τρόικα λαμβάνει μια πολιτική απόφαση. Όταν η ίδια η Επιτροπή ζητάει για μια για 425 εκατομμύρια λέει στην Ευρώπη ότι, στην Ελλάδα συγγνώμη, ότι θα πρέπει να τα πάρετε από τον τομέα της άμυνας λέει ότι θα, δεν θα πάρετε από τον τομέα της άμυνας αλλά από τις ε, μισθούς και τι συντάξει. και όταν εδώ στον ε, Μανουέλ ε, εδώ παίρνει μια πολιτική απόφαση για την Ελλάδα. Πού την έλαβε αυτή την εντολή. Μα εγώ έχω εντολή από το Συμβούλιο, από το ΕΚΟΦΗΝ και τι εκτελώ. Και συχνά λέει, το Συμβούλιο λέει ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην Κομισιόν. Μα εδώ διαλύουμε τη δημοκρατία και παίρνουν αποφάσει πέραν ε, από κάθε ε, λογοδοσία. Ρομπέρτο, δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην ανάγκη μιας πολιτικής ανάπτυξης ε, για την Ελλάδα. Εντάξει, κινητοποίηση των ε, οικονομικών και τεχνικών μέσων, αλλά στην Ελλάδα χρειάζεται μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή ζήτηση. Είπατε ότι δεν θέλετε να επισέλθετε στις λεπτομέρειες και στην ουσία των σχέσεων με, για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα ήθελα όμως να το πράξετε και να μας πείτε τι πιστεύετε για το ότι η Γερμανία με 5,9 ε, πλεόνασμα θεωρείται μια χώρα η οποία δεν ε, δημιουργεί πρόβλημα μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η άλλη ερώτηση είναι μια θεσμική περιέργεια. Το 2PAC είναι μια απόλυτη καινοτομία διότι είναι κανισμή βάσει το 136. Ναι, θα είναι, θα αρμοδιά του, του αλλά θα ψηφίζεται από μόνο από τις χώρες ε, Ευρωζώνης. Λοιπόν, τι ρόλο βλέπετε για το Eurogroup που έχει το έργο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, να ασχοληθεί και ατύπως για ζητήματα τα οποία έχουν ε, σημαντικές επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. Ε, ποιο ρόλο λοιπόν μπορεί να έχει το, Eurogroup στην συζήτηση περί του ΠΑΚ. Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω πρώτα στο Φιλίπ με καλεί να συζητήσω ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν θα το κάνει γιατί θα πρέπει να εκφράσω πάρα πολλές αμφιβολίες. Πολλές αμφιβολίες και πολλά ερωτηματικά. Και δεν θέλω να περιπλέξω το έργο κάποιον και ούτε το δικό μου μαζοχιστής δεν είμαι αλλά θα πρέπει σοβαρά να σας πω ότι η κατανομή της εργασίας υπάρχει και οι ευθύνε επίσης στους διάφορα, στους διάφορους τομείς της ε, Τρόικα. Δηλαδή όπου επίσης το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο κλπ. Το Eurogroup ε, δεν είναι έτοιμο με τις Τρόικας. Εγώ άκουσα έναν επίτροπο που εξηγούσε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα σας πω, ποιος ήταν, υπάρχουν πολλοί, ότι το Eurogroup επέβαλε τη μείωση των, κοινωνικών, των κοινωνικών μισθών. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και εγώ οπωσδήποτε όχι και έχω και μάρτυρες οι οποίοι δεν πρέπει να αφήσουν. Πολλές φορές έκανα ό,τι μπορούσα για να αποφευχθεί η παρέμβαση στους ελάχιστους μισθούς. αλλά κυρίως οι χώρες, και τους καταλαβαίνω κάπως, που έχουν χαμηλότερους ελαχίστους μισθούς από την Ελλάδα, που, το λέω προς Έλληνες φίλος αυτό, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν στα δεκάτα τα συνδικάτα, στους δικό τους κοινή γνώμη, ότι θα πρέπει να διαθέσουν σημαντικότατα ποσά για να βοηθήσουν την Ελλάδα, ενώ εκείνοι έχουν πολύ πολύ χαμηλότερους κοινωνικούς ελάχιστους μισθούς από εκείνους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά δεν συζητάμε στην πολιτική τις λεπτομέρειες των μέτρων που επιβάλλονται σε κάποιους. Ε, για μένα αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Ε, νομιμοποίησης, δημοκρατίας ή το Eurogroup δέχεται τα μέτρα που προτείνει η Τρόικα. Αλλά αν έκανε το Ευρωγκουπ ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που κάνει η Τρόικα, το δούνιο θα απομακρύνεται από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων και αν το δονητού δεν ήταν τμήμα, τότε ορισμένες χώρες δεν θα υποστήριζαν ε, το σύνολο των μέτρων γιατί επιμένουν στην παρουσία και συνοδεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι πραγματικό αυτό το ερώτημα που ε, υπέβαλες και θα ήθελα να μπορούσαμε να το συζητήσουμε μεταξύ δημοκρατών. Ιδίως όσον αφορά τη μείωση του ε, δημοσιονομικού ελλείμματος για αυτά τα 325 εκατομμύρια ε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα, μήνυμα, ένα τμήμα μείωσης των στρατιωτικών ε, δαπανών. Εγώ δεν ήμουν ποτέ παρόντα, παρόν σε μια συζήτηση όπου κάποιος είπε αφήστε τους στρατιωτικούς, τους στρατιωτικούς στη ρησυχία τους, πάτε τα λεφτά που σας χρειάζονται από τους δοξιούχους. Ποτέ δεν ήμουν παρόν σε κάτι τέτοιο. και πραγματικά εγώ θα μπορούσα να ε, συστήσω σε εκείνους που ήταν επί τόπου να εξετάσουν το θέμα των ε, αμυντικών δαπανών. Το βρίσκω σκανδαλώδες που δεν μειώνονται περισσότερο αυτές οι χώρες. Ότι οι άλλες χώρες δεν σταματάνε τις εξαγωγές οπλισμών προς την Ελλάδα. Ε, je εγώ δεν είπα ότι δεν, θέλουμε κάποια, θέλω κάποια στιγμή να συζητήσουμε τους δύο κανονισμούς αυτούς για τις δύο εκθέσεις ε, που έχω τους ε, εισηγητές απέναντί μου. Εγώ απλώς δεν θέλησα να μπω σε λεπτομέρειες σήμερα και δεν θέλησα να σχολιάσω το πλεόνισμα που έχει η Ελλάδα όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, γιατί τότε θα έπρεπε να εξηγήσω γιατί η Γερμανία είναι στο 5,9 ε, το Λουξεμβούργο στο 6,5 δεν ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση τώρα. Είναι πάντως μια συζήτηση σοβαρή που δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Και όχι με απλά ε, επιχειρήματα. Το Eurogroup προφανώς θα παίξει το ρόλο του στη συζήτηση για τις ανοσορροπίες εφόσον τα κράτη-μέλη της ζώνης ευρώ αφορούν από το θέμα Δεν έχουμε ξεκινήσει συζήτηση, θα το κάνουμε 12 και 13 Μαρτίου. Και προφανώς θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα. Η πρόταση εκτός μικροφώνου. Κατάλαβα την ε, απάντηση για τις δύο μας ερώτησεις για την ανισορροπία του ισοζυγίου και το δεύτερο κατά πόσο το Ευρωγκρουπ θα έχει ένα ρόλο στη διαπραγματεύσεις για το Tupac. Και ε, εκεί επίσης πήρα εν μέρη μια απάντηση. Εγώ ικανοποιήθηκα πάντως, Πρόεδρε. So we, we're happy to leave it. Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάτι σπάνιο την επόμενη εβδομάδα, δεν συνεδριάζει η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Η επόμενη συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα 12 Μαρτίου στο Στρασβούργο. λοιπόν.